Uh, θα ξεκινήσουμε. Να σας ενημερώσω ότι υπάρχει απευθείας μετάδοση στο τηλεοπτικό κανάλι του διαδικτύου. Έχουμε μαζί μας τον Γιωχάνες Χάν, τον Επίτροπο, θα του δώσω το λόγο, αλλά θα ήθελα να κάνω κάποιες μικρές ανακοινώσεις. Καταρχάς, ημερήσια διάταξη. Το σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης, της κυρίας Κράτσα δηλαδή, έχει αποσυρθεί μετά από αίτημά της. Και θα συζητηθεί τον μήνα Ιούνιο, στην 3η Ιουνίου, στις 3 συγγνώμη Ιουνίου. Δεν υπάρχει κάποια αίτηση αλλαγής άλλη, μπορεί να θεωρηθεί δεκτή ημερήσια διάταξη. Ένα δεύτερο σημείο, αφορά τα πρακτικά των τελευταίων συνεδριάσεων της 17ης και 18ης Μαρτίου. Είναι διαθέσιμα τα πρακτικά αυτά, έχουν διορθωθεί, έχουν διανεμηθεί και θα θεωρηθούν δεκτά στο τέλος της συνεδρίασης εφόσον δεν εκφραστεί αντίρρηση από πλευρά σας. Τρίτο σημείο. Οι προσωπικές ανακοινώσεις του Προέδρου, αν θέλετε. Ενθυμίστε ότι είχαμε πάρει μια απόφαση τον μήνα Σεπτέμβριο να αποστείλουμε μια αντιπροσωπεία στην περιοχή του Παρισίου, των Παρισίων. Θα υπάρξουν δέκα συνάδελφοι που θα πάνε από την Επιτροπή μας. Οι τέσσερις θα είναι Γάλλοι. Στόχος είναι να δουν επιτόπου πώς εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκές πολιτικές στα πλαίσια των γαλλικών πόλεων. Οπότε τώρα περνάω στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Ανταλλαγή απόψεων με τον Γιωχάνες Χάν, τον υπεύθυνο για την περιφερειακή πολιτική. Έχετε την ελευθερία κύριε Επίτροπε να μας παρουσιάσετε ό,τι ε, θεωρείτε σχετικό με την πολιτική συνοχής. Ευχαριστώ Ντανούτα. Κύριε και κύριοι, χαίρομαι πολύ που για πρώτη φορά σήμερα θα συζητήσω μαζί σας εδώ ε, και αναμένω πως ε, θα υπάρξουν πολλές ακόμα συναντήσεις που θα διαδεχτούν τη σημερινή. Ε, όπως είναι γνωστό, βρισκόμαστε στο ίμιση περίπου της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου και στο τέλος αυτής της περίοδου πάνω από 2 εκατομμύρια projects θα έχουν υλοποιηθεί, 2 εκατομμύρια τρόποι για να καταστεί ορατή η Ευρώπη για τους ε, πολίτες, τους και τις, α, τους πολίτες και τις πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω πως είναι ε, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία ώστε να ενισχυθεί η το θετικό αίσθημα για την Ευρώπη σε μια περίοδο που πολλοί θεωρούν πως η Ευρώπη υπάρχει μόνο για να προβαίνει σε ελέγχους ε, και να συνιστά περικοπές. Θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα ότι η Ευρώπη υπάρχει και για να αναπτύξει τις ε, περιφέρειες και να δώσει νέες προοπτικές στους ανθρώπους. Αυτό είναι το δικό μας καθήκον και είχα ήδη πει πως δεν υπάρχει κάποια άλλη αναλλακτική απέναντι στην ε, περιφερειακή πολιτική. Πέρα από μια ακόμα καλύτερη ε, και πιο φιλική προς τις μεταρρυθμίσεις περιφερειακή πολιτική. Και γι' αυτό θα πρέπει να αξιοποιήσουμε και το τρέχον έτος, το 2010, το οποίο είναι καθοριστικό και για την ε, μελλοντική διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής, εν ώψη και της Στατικής 2020 και των συζητήσεων που βασίζονται και σχετίζονται με αυτή σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό και την αναθεώρηση του προπολογισμού. Ε, πριν από μερικές ημέρες είχαμε την έκθεση, τη συνδετική έκθεση σε ό,τι αφορά την ε, προγραμματική περίοδο 2000-2006 και είδαμε εκεί πως υπάρχουν κάποια πολύ σημαντικά και πολύ απτά αποτελέσματα όπως για παράδειγμα η δημιουργία τεσσάρων εκατομμυρίων θέσεων εργασίας ή το γεγονός ότι 20,5 εκατομμύρια πολίτες εποφελούνται πλέον τώρα από συστήματα καθαρισμού των αποβλήτων των υγρών αποβλήτων, πράγμα το οποίο ε, συμβάλλει στην ακόμα καλύτερη υγιεινή. Προφανώς ε, δεν έχουν τελειώσει τα καθήκοντά μας, υπάρχουν ακόμα προβλήματα τα οποία καλούμαστε να επιλύσουμε. Είδαμε πως ε, γίνονται όλο και περισσότερες επενδύσεις στον χώρο της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας αλλά και έχουμε και έναν τριπλασιασμό των σχετικών κοντιλίων σε ό,τι αφορά την έρευνα και την καινοτομία σε σύγκριση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο ενώ δίνεται ταυτόχρονα και ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην αξιολόγηση και στην εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγηση εξάντε και εξπός. Θα ήθελα τώρα να σας ενημερώσω σε σχέση με κάποιες τρέχουσες εξελίξεις και προφανώς ε, να δώσουμε ε, εδώ την ευκαιρία και να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που μας δίνεται για ανταλλαγή απόψεων. Πριν από μερικέ εβδομάδε, νομίζω ότι μεγάλη εβδομάδα είμαστε σε, ε, σε θέση να παρουσιάσουμε τη νέα στρατηγική έκθεση για μια πολιτική συνοχή που θα, που θα βασίζεται και θα στοχεύει σε ακόμα περισσότερη απόδοση και είχαμε τη δυνατότητα μια από κοινού έκθεση έκθεσης σε ό,τι αφορά τα, τους μα μας ε, στόχους για τη κοινή διαχείριση συνεπάγεται και κοινή ανάληψη ευθύνης. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τα κράτη-μέλη για την ε, συνεισφορά τους ε, στη σύνταξη αυτής της έκθεσης γιατί κάτι τέτοιο θα αποτελέσει τη βάση για την σύνταξη αντίστοιχων εκθέσεων αλλά και για τη λήψη αντίστοιχων μέτρων που θα ενισχύουν και θα εκφράζουν την ανάληψη της δέσμευσης από την πλευρά των κρατών μελών για μια τέτοια πολιτική. Είδαμε ότι χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια και μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στους ε, πολίτες της ε, Ευρώπης. Ποια είναι λοιπόν τα συμπεράσματα και οι συστάσεις ε, για το μέλλον. Ας ξεκινήσουμε με, τα, με τις θετικές συστάσεις και τα συμπεράσματα. Συνολικά λοιπόν τα κράτη-μέλη καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες ε, τόσο στο επίπεδο της υλοποίησης των ε, προγραμμάτων αλλά και στο πλαίσιο της ε, επιλογής και στο πλαίσιο της χρηματοδότησης. Σε αυτή τη φάση έχουν ήδη διατεθεί 93 δισεκατομμύρια ευρώ για αντίστοιχα προγράμματα, δηλαδή βρισκόμαστε γύρω στο 27% του συνολικού προπολογισμού, με βάση βέβαια ε, την οικονομική ε, κρίση. Ε, αντιλαμβάνεστε πως η χρηματοδότηση από την πλευρά των κρατών μελών αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία. Γιατί δεν βρισκόμαστε ακριβώς στο ίδιο επίπεδο η χρηματοδότηση έχει κινηθεί στα ίδια επίπεδα όπως και κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και ήδη από 14 κάτι μέλη μας ε, ανέφεραν ότι συνολικά έχουν δημιουργηθεί 350.000 ε, νέες θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να αναφερθούμε και στα σημεία κριτικής, στα αρνητικά ζητήματα. Διαπιστώσαμε ε, πως υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά την υλοποίηση προγραμμάτων σε ορισμένους τομείς, ειδικότερα στον τομέα της ενέργειας, στην υλοποίηση των ευρυζωνικών δικτύων αλλά και στον περιβαλλοντικό τομέα και σε ό,τι αφορά τέλος και τις δυνατότητες διοίκησης, δηλαδή τις υποδομές διοίκησης. Και να πούμε εδώ πως αυτές οι καθυστερήσεις ε, συχνά δεν οφείλονται σε ζητήματα χρηματοδότησης αλλά σε άλλα, ε, σε άλλους ε, λόγους. Για παράδειγμα, όπως είδαμε και στον χώρο του περιβάλλοντος, υπάρχουν διατάξεις κοινοτικέ οι οποίες δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών και κατά συνέπεια δεν υπάρχει απαραίτητη νομική βάση για την λήψη μιας χρηματοδότησης κοινοτική. Δηλαδή, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα μεγαλύτερα προγράμματα, χρειαζόμαστε να έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή σχετικέ νομικέ διατάξεις και αυτό θα πρέπει να διασφαλιστεί. Και ακριβώ γι' αυτό σα καλώ και εσά από τη δική σας πλευρά να κάνετε τις κατάλληλες προσπάθειες σε συνεννόηση με τους ε, εθνικούς σας συναδέλφους. Επίσης υπάρχει μια συμμετρία ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την επιλογή των ε, projects, των προγραμμάτων. Και από την άλλη πλευρά θα ήθελα να τονίσω πως αυτή η στρατηγική έκθεση αποτελεί ένα είδος συνάψεων, δηλαδή ε, μια απεικόνηση της κατάστασης όπως έχει αυτή τη στιγμή. Και είδαμε πως ε, και από τις εθνικές αξιολογήσεις ε, υπήρχε κάποιος εκνευρισμός ή κάποια δυσαρέσκεια σε πολιτικό επίπεδο ως προς το τι λαμβάνεται ή δεν λαμβάνεται υπόψη. Αλλά συνολικά το συμπέρασμα είναι σωστό αυτή τη έκθεση. Όμως θα πρέπει να αναφέρουμε πως ε, κράτη-μέλη βασίστηκαν ε, στην περίοδο από το αρχές Ιουνίου στα τέλη Νοεμβρίου ή Δεκεμβρίου ε, με αποτέλεσμα να υπάρχει η, βασική, η συνολική εικόνα που έχουμε να μην είναι ακριβώς αντίστοιχη μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά δηλαδή την απορρόφηση των κονδυλίων. Γιατί ε, ειδικά σε ό,τι αφορά την ε, πρώτη περίοδο, τον πρώτο μισό χρόνο για παράδειγμα της προγραμματικής περίοδου, συχνά λαμβάνουν χώρα πολλές σημαντικές αλλαγές σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να καλέσω τα κράτη-μέλη να προωθήσουν περαιτέρω την υλοποίηση, ούτως ώστε τα κονδύλια που έχουν διατεθεί να μπορέσουν πράγματι να αξιοποιηθούν. Ε, νομίζω πως ε, ε, όλοι εδώ συμφωνούμε πως ο στόχος της περιφερειακής πολιτικής δεν μπορεί να είναι η εξοικονόμηση των εισαγωγικών πόρων. Ο στόχος πρέπει να είναι η σωστή, η αποτελεσματική και η βιώσιμη αξιοποίηση αυτών των πόρων, μια βιώσιμη τέτοια περιφερειακή πολιτική, ούτως ώστε να μπορούμε στο τέλο τη προγραμματική περίοδου όχι ήμασταν σε θέση να εξοικονομήσουμε πόρους αλλά αντίθετα ήμασταν σε θέση να αξιοποιήσουμε αυτούς τους ε, πόρους ε, υλοποιώντα επιτυχή και βιώσιμα έργα. Νομίζω πως και στο μέλλον θα είναι σημαντικό η συγχρηματοδότηση να συνεχίσει να εκφράζει ακριβώς την ανάληψη τη δέσμευσης από την πλευρά των κρατών μελών ως βασική αρχή και θεωρώ πως ειδικότερα η επένδυση σε πρωτοβουλίες περιφερειακής πολιτικής αποτελεί κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό για την οικονομική ανάκαμψη. Τώρα, ε, πώς θα συμβάλλει η περιφερειακή πολιτική στρατηγική 2020. Σίγουρα θα πρέπει η περιφερειακή πολιτική να προσαρμοστεί στις τρέχουσες εξελίξεις. Τα αποτελέσματα όμως ε, στα οποία αναφερθήκα εν το πόσο σημαντικό είναι αυτό το εργαλείο της περιφερειακής πολιτικής για την ανάπτυξη και την απασχόληση και κατά συνέπεια η πολιτική συνοχή θα πρέπει να τεθεί στην υπηρεσία της στρατηγικής 2020. Εάν θέλουμε ανάπτυξη η οποία θα είναι έξυπνη, θα είναι πράσινη και ολοκληρωμένη, χρειαζόμαστε όμως ταυτόχρονα ε, και την ε, δέσμευση των ε, κατάλληλων πόρων και η πολιτική συνοχή μας δίνει το κατάλληλο πλαίσιο στους εκάστοτε τομείς αλλά και σε συγκεκριμένες περιφέρειες να προτείνουμε λύσεις λαμβάνοντας υπόψη και την Ευρωπαϊκή Συνοχή. Η περιφερειακή πολιτική έτσι όπως τη φανταζόμαστε από κοινού και αυτό μπορούμε να το επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι γίνονται οι κατάλληλες επενδύσεις πόρων στις περιφέρειες. Και θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ξανά και ξανά τον όρο αυτό, την επένδυση. Όχι το sponsoring, τη χρηματοδότηση ή την χορήγηση, αν θέλετε, ενισχύσεων αλλά να χρησιμοποιούμε τον όρο επένδυση, γιατί το επένδυση σημαίνει ότι θα υπάρξει απόδοση από αυτή την επένδυση, θα υπάρξει return αυτό που λέμε. Μπορούμε βέβαια να μιλήσουμε για το τι είδος return ακριβώς αναμένουμε από μια επένδυση, αλλά αυτό που θα πρέπει να ισχύει είναι ότι χρειάζεται μια αντίστοιχη και νέα ανάπτυξη των ε, περιφερειών, ώστε να μπορέσει αυτή η πολιτική να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα να συμβάλλει και στην ε, καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών της Ευρώπης. Αυτό όμως που χρειαζόμαστε, και το ξαναείπα ταυτόχρονα, είναι η η εστίαση σε ορισμένες λίγες προτεραιότητες αφενός, αλλά αφετέρου και μια μέγιστη ευελιξία σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των διαφόρων προγραμμάτων στις 270 ε, διαφορετικές περιφέρειες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, διαπιστώνουμε ότι 230 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν δεσμευτεί στο πλαίσιο της πολιτικής της Λισαβόνας. Και από αυτά 86 ε, δισεκατομμύρια ε, για την έρευνα και την καινοτομία, ε, 48 ε, δισεκατομμύρια σε ό,τι αφορά τις κλιματικές μεταβολές, την, πιο φιλοπεριβαλλοντικές μεταφορές και το τομέα της ενέργειας. Όμως, και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε για μία ακόμα φορά, χρειάζεται η μέγιστη ευελιξία στο επίπεδο της υλοποίησης. Και εδώ θα πρέπει να βασιστούμε στις αδυναμίες αλλά και στα προσόντα τις εκάστοτε περιφέρειες. Εκείνο που δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να κάνουμε είναι να έχουμε ε, μια ταυτότητα USP, ε, δηλαδή ε, ένα χαρακτηριστικό το οποίο θα αφορά ακριβώς τις ιδιαιτερότητες μιας περιφέρειας ώστε να μπορούν οι επενδύσεις που θα γίνονται να βασίζονται στα δυνατά στοιχεία της εκάστοτε περιφέρειας. Και νομίζω πως αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν βρισκόμαστε εν μέσω της συζήτησης για τη στρατηγική 2020. Ε, Και εδώ σας ε, καλώ στις δικές σας ε, εκλογικέ περιφέρειες, στις συζητήσεις που γίνονται στο εθνικό επίπεδο στα κράτη-μέλη σας, να τονίζετε ότι όταν υπάρχουν ευρωπαϊκοί στόχοι, μιλάμε για στόχους ευρωπαϊκούς με βάση μέσους όρους και σας λέω ότι ξέρω ότι γνωρίζω αυτά τα πράγματα γιατί όταν μιλάμε για αυτό το στόχο του 3% γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποια, α, κάποιες ε, περιφέρειες και κάποια μέλη τα οποία βρίσκονται πολύ πιο πάνω από αυτό το 3% και κάποια πολύ πιο κάτω. Άρα λοιπόν θα πρέπει πέρα από τα, ε, τους ευρωπαϊκούς στόχους να έχουμε και εθνικούς στόχους οι οποίοι θα είναι φιλόδοξοι και οι οποίοι στο σύνολό τους τελικά θα ανταποκρίνονται σε αυτούς τους συνολικούς ευρωπαϊκούς στόχους. Άρα λοιπόν ένα από τα σημαντικά συμπεράσματα τα οποία θα πρέπει να λύσουμε από την Λισαβόνα είναι ακριβώς η μεταφορά αν θέλετε η μετάφραση των συνολικών ευρωπαϊκών στόχων σε συγκεκριμένους εθνικούς στόχους. Γιατί ε, όταν λέμε για ένα συγκεκριμένο στόχο ότι κάποιοι θεωρούν πως ένα τέτοιο στόχος είναι υπερβολικά φιλόδοξος ενώ κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι είναι πολύ χαμηλός ε, το καλύτερο σε αυτή την περίπτωση είναι να έχουμε συγκεκριμένους ε, στόχους ούτως ώστε ε, να διασφαλίσουμε με πολύ καλύτερο τρόπο ότι η στρατηγική 2020 θα εφαρμοστεί με τον κατάλληλο τρόπο. τελικά αυτό που είναι το ζήτημα εδώ είναι η διαχείριση της κρίσης, το κλείσιμο των σχετικών κενών και το να αποτρέψουμε τα να δημιουργηθούν μεγαλύτερα κενά από αυτά που υπάρχουν ήδη, ούτως ώστε να μπορέσει να διατηρηθεί όσο έχει το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Ε, ταυτόχρονα σύντομα μέσα από μερικέ εβδομάδε θα παρουσιαστεί και η πέμπτη, πέμπτη έκθεση σε ό,τι αφορά το μοντέλο για τη συνοχή και εκεί θα υπάρχουν συγκεκριμένε προτάσει για την όλη συζήτηση και για μένα ήταν σημαντικό αυτή η έκθεση να περιληφθεί και μέσα στις ε, πρωτοβουλίες ε, του ε, προγράμματος εργασιών, της εργασιών Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκεί λοιπόν περιλαμβάνεται μια σημαντική ενίσχυση πλέον της πολιτικής συνοχής ως συνολικός στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμπληρωματικά πριν από το καλοκαίρι κάπου τον Ιούλιο δηλαδή από άποψη εποχών μέσα στο καλοκαίρι, αλλά και μετά από τι κανονικέ διακοπέ, θα έχουμε δύο ανακοινώσει ό,τι αφορά την καινοτομία και την βιωσιμότητα, όπου θα απευθυνθώ ε, και έχω ήδη καλέσει άλλους ε, επιτρόπους ε, και τις γενικές διευθύνσεις να συμμετάσχουν στην εκπόνηση αυτών των εκθέσεων ώστε να έχουμε μια συνεκτική, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε ό,τι αφορά αυτά τα συστήματα. Ε, τέλος, επιτρέψτε να κάνω μια παρατήρηση σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του προϋπολογισμού. τα καθήκοντα της περιφερειακής πολιτικής δεν έγιναν λιγότερα. Αντίθετα, δεν θα αποτελέσει έκπληξη για εσά, ούτε για μένα αποτελεί έκπληξη και νομίζω πω ήταν ούτε αυτό το γνωρίζει καλά. Κατά τη διάρκεια των εβδομάδων ε, της δικής μου θητείας, ε, ήδη ε, υπήρξε ένα ένας κατάλογο κατάλογος επιθυμιών ε, που μου προτάθηκαν διάφορες πρωτοβουλίες, διάφορα νέα μέτρα και προγράμματα και γνωρίζουμε πως μια λογική, μια σωστή περιφερειακή πολιτική δεν μπορεί να γίνει με μηδενικό κόστο. Χρειαζόμαστε τον κατάλληλο προπολογισμό, τα κατάλληλα κονδύλια. Το λέω πολύ ανοιχτά. Εάν ο συνολικός προπολογισμό δεν ε, φτάνει ένα σημαντικό μέγεθος, τότε όλα αυτά τα σημαντικά projects, όλα αυτά τα έργα τα οποία οραματιζόμαστε και τα οποία θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο, θα είναι δύσκολο να εφαρμοστούν. Άρα, είναι σημαντικό και εδώ σας καλώ τόσο εντός του ε, Κοινοβουλίου αλλά και εντός των ίδιων των πολιτικών ομάδων να ε, προωθήσετε την ιδέα της καλύτερης ενσωμάτωσης των διάφορων τομεακών πολιτικών στην περιφερειακή πολιτική, ούτως ώστε να μην λάβει χώρα ένας του προϋπολογισμού. Ε, πέρα όμως από αυτή τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, θα πρέπει να μας απασχολήσουν και τα νέα ε, μοντέλα χρηματοδότησης. Ε, λαμβάνει η χώρα μία αν θέλετε μεταμόρφωση, μία αλλαγή σε ό,τι αφορά την κουλτούρα που ακολουθούμε. Γιατί εάν στο πλαίσιο αυτής της λογικής που λέγαμε τη επένδυσης, ε, ότι δηλαδή θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η απόδοση, προφανώς θα είναι ε, σημαντικό κανείς εκ των προτέρων να ε, εξετάζει το αν μια τέτοια επένδυση είναι λογική, έχει νόημα σε αντίθεση με την χορήγηση μια απλής ενίσχυση επιδότηση. Έτσι ε, μια τέτοια προσέγγιση ε, θα, νομίζω πως θα οδηγήσει σε υψηλότερα ποσοστά επιτυχία σε ό,τι αφορά τα έργα μας και ταυτόχρονα ε, μια τέτοια προσέγγιση θα μας βοηθάει να αποφεύγουμε λάθη και να σας πω ότι έχει συσταθεί μια ομάδα εργασίας μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Μάρκ και Γενικής Διεύθυνσης Regio σε ό,τι αφορά το public procurement, δηλαδή την, το μέτρο δημόσιων προμηθειών. Και μιλάμε εδώ για δύο μεγάλους τομείς οι οποίοι ευθύνονται για υψηλά ποσοστά στον των χωρίς όμως να, εμείς να έχουμε να παίξουμε μεγάλο ρόλο εδώ. Οπότε αν μπορέσουμε να λάβουμε καλύτερα υπόψη μας τις ε, ανάγκες ε, που υπάρχουν στο πλαίσιο των, της ε, ανάθεσης ε, τέτοιων ε, δημόσιας ανάθεσης ε, έργων νομίζω πως θα οδηγηθούμε και σε, μια καλύτερη, σε ένα καλύτερο σχεδιασμό αλλά και αξιοποίηση της, των διάφορων διαθροτικών κοντιλίων και έχοντα κάνει αυτά τα σχόλια θα κλείσω εδώ και αναμένω τη συζήτησή μας. I think... Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Μπορούμε τώρα να αρχίσουμε τη συζήτηση είστε να αρχίζουμε με τους συντονιστές, αλλά δεν εκδήλωσαν ε, συντονιστές ε, ιδιαίτερα ενδιαφέρον να μιλήσουν. Ο κύριος Λαμπέρτ ε, Βανίστελ Ρόι. Eh, eh, Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα, κύριε Επίτροπε, να σας ευχαριστήσω καταρχήν για την ενημέρωση που μας κάνατε. Θα προσπαθήσω να είμαι λακωνικός. Ήταν πολύ θετικές εντυπώσεις που μας αφήσατε στην ακρόασή σας. Και ήταν πολύ εμπεριστατωμένες οι πληροφορίες που μας ε, δώσατε. Έχω μερικές ερωτήσεις όμως. Ποια είναι η γνώμη σας ε, για την ενδιάμεση αναθεώρηση των ε, χρηματοπιστωτικών θεμάτων και των δημοσιονομικών ε, προοπτικών. Εσείς θα συμμετάσχετε σε αυτή την ενδιάμεση αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών. Δεν ξέρω ε, αν αυτό είναι κάτι καλύτερο από έναν επίσημο έγγραφο ή θα πρέπει να περιμένουμε πρώτα την έκθεση της συνοχής για να αξιολογήσουμε το έργο που έχει γίνει μέχρι τώρα. Και δεν ξέρω τι έχετε συμφωνήσει με τον κύριο Μπαρόζο. Μιλήσατε και για τις μακροπεριφέρειες. Το είχατε αναφέρει και στην ακρόαση. Θα ήθελα όμως να αναπτύξετε λίγο περισσότερο αν γίνεται τα κριτήρια. Με βάση ποια κριτήρια θα εφαρμοστεί αυτό το νέο μόρφωμα στην Ευρώπη. Επίσης, ε, για την περιοχή του Δούναβη. Αργότερα θα, στο έτος θα πραγματοποιήσουμε και αποστολή στην περιοχή αυτή. Γι' αυτό θα ήθελα κάποια στοιχεία. Αυτά προς το παρόν. Thank Η κυρία Κρέλ. Äh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, έχω τρία ερωτήματα τα οποία θα ήθελα να σας θέσω ε, και σε σχέση με το midterm review. Ε, στο παρελθόν λοιπόν είχαμε θέσει επανειλημμένα αυτό το ερώτημα του κατά πόσο θα πρέπει ε, να επενδύσουμε κονδύλια από αυτό το τομέα στο κατασκευαστικό τομέα για τις ε, κατοικίε, ε, ε, Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο έχετε στοιχεία για το πώς γίνεται η υλοποίηση σε αυτό το επίπεδο από την πλευρά των κρατών μελών και το αν υπάρχει υλοποίηση ή αν υπάρχει αυτό τελικά αναλώνεται μόνο σε wishful thinking, δηλαδή απλά και μόνο σε σχετικέ επιθυμίε, αλλά τίποτα στην πράξη. Μετά, εδώ το Κοινοβούλιο θεωρεί πως τα κονδύλια τα οποία ενδεχομένω δεν θα δαπανώνται στο επίπεδο των n 2 και n 3 να διατηρούνται για άλλα διαρθρωτικά έργα και άλλους ε, τομείς χωρίς δηλαδή να επιστρέφονται αυτά τα κονδύλια στα κράτη-μέλη. Ποια είναι η δική σας ε, ε, θέση. Θα μπορούσε δηλαδή να συγκεντρώσει μια τέτοια θέση την πλειοψηφία των κρατομελών στο Συμβούλιο, ώστε σε ό,τι αφορά την στρατηγική του Δούναβη ή τη ε, βαλτική Οδό, ώστε να μπορέσουν αυτά τα κονδύλια να διατηρηθούν για να ε, επενδυθούν σε άλλα αντίστοιχα έργα. Ε, και μια τρίτη ερώτηση. Υπάρχουν κάποια στοιχεία σχετικά με την ε, ροή των κοντιλίων τα οποία από την πλευρά της περιφερειακής πολιτικής ε, μπορεί να έχουν συμβάλει στην ανάκαμψη από την οικονομική κρίση. Δηλαδή για να έχουμε αν θέλετε μια ιδέα ως προς το κατά πόσο πράγματι η περιφερειακή πολιτική μπορεί να βοηθήσει στην πραγματικότητα τα επιμέρους κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε μία ακόμη ερώτηση και μετά θα δώσουμε το λόγο στον Επιτροπό κύριο Μάνα Μανέσκου. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν κύριε Επίτροπε να σας συγχαρώ για το ότι αναγνωρίσατε τη σημασία που έχει η ανάμειξη των εθνικών και περιφερειακών αρχών στην περιφερειακή πολιτική. Και ελπίζω την ίδια διαλεκτικότητα να δείξετε απέναντι σε εθνικές και περιφερειακές αρχές ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για το πρόγραμμα Έρασμος. για τους εκπροσώπους των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Στην έκθεση πρωτοβουλίας μου επισήμανα την ανάγκη συνέχισης του προγράμματος Έρασμος και για τους εκπροσώπους των Δήμων και Κοινοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντίθετα είπε ότι θα διακόψει αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Ερωτώ λοιπόν κύριε Επιτροπέ, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε αυτή την απόφαση διακοπής του προγράμματος και επίσης ε, θα ήθελα πιο διεξοδικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τα αρνητικά αποτελέσματα των μελετών ε, σκοπιμότητας που έγιναν. Η δεύτερη μου ερώτηση αφορά την δημοσιονομική αναθεώρηση και το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτό το θέμα που εξετάστηκε πέρυσι. Έγιναν κάποιες προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατανομή των κονδυλίων και την κατάργηση του στόχου 2 ή τον περιορισμό της χρηματοδότησης σε μια συγκεκριμένη περίοδο πεπερασμένη μετά τη διεύρυνση. Τέτοια μέτρα είναι απαράδεκτα ε, για πολλά νέα κράτη-μέλη. Ποια είναι η δική σας γνώμη για τις προτάσεις αυτές. Πότε αναμένετε το επίσημο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοσιονομική Αναθεώρηση και τη θέση της πολιτικής συνοχής στο νέο σχέδιο προϋπολογισμού. Thank you. So we would... Ωραία, τώρα θα δώσουμε το λόγο στον Επίτροπο για να σχολιάσει και να απαντήσει στις ερωτήσεις. Yeah, Ευχαριστώ καταρχήν σε ό,τι αφορά το όλο οικονομικό ζήτημα. Νομίζω πως το τρίτο τρίμηνο ή εν πάση περιπτώσει μετά το καλοκαίρι, δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, να δημοσιευθεί αυτό το budgetary midterm review, η ενδιάμεση δηλαδή έκθεση αναθεώρησης για τον προπολογισμό και ειδικότερα η περιφερειακή, η πολιτική ως ένας από τους Big Spender, δηλαδή από τους τομεί που έχουν μεγάλου ε, προπολογισμού θα απασχολήσουν εδώ αυτή την έκθεση με μια αντίστοιχη ομάδα εργασίας και προφανώς εμείς έχουμε μπλακεί στην ε, στο, στο να καταγράψουμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Από εκεί και μετά, σε ό,τι αφορά τις μακροπεριφέρειες. Να συνοψίσω. Ε, υπάρχουν τα τρία εννοώ. Δύο εκ των οποίων είναι ας πούμε συμπαθητικά και το τρίτο δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι συμπαθητικό, αλλά εν πάση περιπτώσει σε ό,τι αφορά τα δύο πρώτα νότα, θα γνωρίζετε, σε ό,τι αφορά δηλαδή ε, έλλειψη αντίστοιχων ε, οργανισμών αυτοδίκης και ούτω καθεξής και το τρίτο είναι η ε, έλλειψη κοντιλίων. Σε ό,τι αφορά τη στατική που αναφερθήκατε, σε ό,τι αφορά την πολιτική στο Ντούναβι ή την πολιτική στη Βαλτική, τα ασιατικά προγράμματα εδώ υλοποιήθηκαν ε, με χρηματοδότηση από τα αντίστοιχα ταμεία γειτονία, αλλά σε ό,τι αφορά την πολιτική ε, Δούναβη, στην περιοχή του Δούναβη ε, και μέσω των μηχανισμών για την χρηματοδότηση των υποψήφιων χωρών. Άρα λοιπόν, ναι, υπάρχουν μια σειρά από ιδέε και προγράμματα σε σχέση με συγκεκριμένες περιφέρειες, αλλά εκεί μπορούμε να συνδυάσουμε με καλύτερο τρόπο τι επιμέρους αυτές τις ιδέες και πρωτοβουλίε. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά έργα ε, τα οποία απαιτούν την ταυτόχρονη συνεισφορά διαφορετικών περιφερειών και ταυτόχρονη υλοποίηση έχουμε ήδη εδώ μια μεγαλύτερη προσθέμενη αξία. Για παράδειγμα, θα σας αναφέρω κάποια παραδείγματα. Ε, σε ό,τι αφορά την, ε, το Δούναβε. Ε, και έχουμε κάποιες μία υποδομή σε ό,τι αφορά τον καθαρισμό των υδάτων σε ένα συγκεκριμένο σημείο κατά μήκο του ποταμού και λίγο πιο κάτω υπάρχει πάλι κάτι το οποίο κάποια έξοδος αποβλήτων προφανώς δεν έχει κάτι τέτοιο νόημα δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία ή για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τους αυτοκινητόδρομους. Ε, δεν έχει νόημα να, ένας αυτοκινητόδρομος να φτάνει μέχρι ε, κάποια σύνορα ε, και μετά, γιατί το έχω ζήσει και αυτό, να, στην, από την άλλη πλευρά των σύνορων στο άλλο κράτος μέλος να μην υπάρχει τίποτα, να μην υπάρχει σχεδόν καθόλου αυτοκινητόδρομος. Άρα λοιπόν αυτό που εννοώ είναι ότι αν χρειάζεται συνεργασία μεταξύ κρατών μελών θα πρέπει να διασφαλίζεται και η συνεργασία μεταξύ τους και η ε, επένδυση των κατάλληλων ε, κοντιλίων, τόσο ώστε ακριβώς να εκμεταλλευόμαστε αυτήν την ε, τη συνέργεια που δημιουργείται. Και σε ό,τι αφορά την αναφορά που γίνεται ότι χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια, απαντώ ότι αξιοποιήστε καταρχήν στο σύνολό τους τα συνολικά διαθέσιμα κονδύλια και θα δούμε από εκεί και μετά. Σε ό,τι αφορά το Δουναβί. Υπάρχουν διάφορες ε, διασκέψεις. Ε, την, ε, στη Βιέννη και στην Πατρισλάβα την προηγούμενη εβδομάδα είχε λάβει χώρα η τρίτη από αυτές τις διασκέψεις. Η επόμενη θα λάβει χώρα στη, στη Βουλγαρία και τον Ιούνιο, η πέμπτη στη Ρουμανία. Και έτσι με βάση αυτές τις διασκέψεις θα έχουμε μία βάση ενώ από το Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο είχε ήδη λάβει η χώρα ε, μια γραπτή διαδικασία διαβούλευσης από την οποία προέκυψαν 70 συγκεκριμένες ε, και σημαντικές ε, τοποθετήσεις. Άρα λοιπόν μέχρι τα τέλη του χρόνου θα έχουμε μια συνεκτική πολιτική η οποία μέχρι το τέλος της επόμενης Προεδρίας θα έχει ολοκληρωθεί θα έχει υλοποιηθεί, θα έχει περάσει το επίπεδο τη υλοποίηση, αλλά θα ήθελα όμω να επαναλάβω και αυτό που είπα και στο πλαίσιο τη διάσκεψη, δηλαδή στι μακροπεριφέρειε ε, γενικά και στη ε, περιφερειακή πολιτική ισχύει η αρχή τη επικουρικότητα. Τι σημαίνει επικουρικότητα, ο καθένα πρέπει να κάνει όσα μπορεί από τη δική του πλευρά και ό,τι δεν μπορεί να το πράξει μόνο του προσφεύγει στο ανώτερο επίπεδο. Αυτό το λέω γιατί έχω την αίσθηση πως ορισμένες περιφέρειες ε, θεωρούν πως μπορούν να επιλύσουν τα προβλήματά τους εάν τα μεταθέσουν, αν θέλετε, ε, στις μακροπεριφέρειες. Αλλά η πολιτική με μακροπεριφέρειες δεν έχει αυτό το στόχο. Ε, μια τέτοια πολιτική μακροπεριφερειών θα πρέπει να αναπτύσσεται μόνο εφόσον ε, υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να επιληθούν στο επίπεδο των επιμέρους περιφερειών. Μία απλή δηλαδή ανάθεση, αν θέλετε, τέτοιο προβλημάτων στο ανώτερο επίπεδο δεν επιλύει κάτι. Ε, σε ό,τι αφορά ε, τον, ε, τα κονδύλια σε ό,τι αφορά κατασκευή κατοικιών, σας λέω δεν ξέρω, δεν έχουμε ακόμα σχετικά στοιχεία. Τώρα σε ό,τι αφορά ε, περιφέρειες N2 ή N3 δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η σχετική περίοδος είχαμε συμφωνήσει στα τρία χρόνια εμείς ούτως ώστε να μην συμβεί τίποτα αλλά με βάση τη στάση σώματος αν θέλετε που βλέπω εδώ από τους ευρωβουλευτές να πούμε πως εδώ ε, δεν σκοπεύουμε να προβούμε σε μια ε, περαιτέρω ε, διεύρυνση. Σε ό,τι αφορά τις προκαταβολές είχαμε 29 δισεκατομμύρια ευρώ συν 6,2 το προηγούμενο έτος. και εάν ε, συμφωνηθεί ε, στο άμεσο μέλλον θα προσθεθούν άλλα 775 εκατομμύρια ευρώ για πέντε κράτη-μέλη, ούτως ώστε να διασφαλιστεί μια συνολική, αν θέλετε, συνεισφορά στη ρευστότητα της τάξης των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ επιπρόσθετα. Ε, σε ό,τι αφορά το, το ζήτημα του προϋπολογισμού δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να προχωρήσουμε είχαμε εξαντλήσει το σχετικό προϋπολογισμό και θα πρέπει να δούμε πώς θα δώσουμε μια συνέχεια γιατί ως προς το στο νόημα ή τη λογική αν θέλετε ενό τέτοιου βήματος ε, προφανώς και συμφωνούμε όλοι ότι δηλαδή χρειάζεται μια τέτοια ανταλλαγή ε, προσώπων, αν θέλετε, πολιτικών προσώπων σε επίπεδο περιφερειών και ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε ε, σε ό,τι αφορά το ζήτημα που αναφέρατε σε ό,τι αφορά το γενικό πλαίσιο της κρίσης, προφανώς αυτό είχε ληφθεί υπόψη και από το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής και η περιφερειακή πολιτική έχει λάβει περισσότερη έμφαση εδώ. Η ευαισθησία, αν θέλετε, ε, αν θέλετε έχει αυξηθεί σε σχέση ε, με αυτό το σημείο και σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε, για τις εξηγήσεις σας. εντυπωσιάζομαι από τη στρέβλωση που παρουσιάζει η παρουσίαση την οποία κάνατε για τις συνθήκες οι οποίες είχαν επικρατήσει στη διαμόρφωση των προγραμμάτων και στη σημερινή κατάσταση. Τα πράγματα διαφέρουν, τα πράγματα έχουν στρεβλωθεί πολύ και δεν ξέρω αν οι ρυθμίσεις τις οποίες προτείνεται μπορούν να καλύψουν τις στρεβλώσεις αυτές αίσθησή μου, λέει ο κ. Αλφονσί, είναι ότι θα πρέπει στα μέσα της διαδικασίας να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε σε βάθος μέτρα για να σκεφτούμε με ποιο τρόπο θα είμαστε αποτελεσματικοί στο μέλλον και να βοηθήσουμε τις περιφέρειες στην ανάπτυξή τους. Υπάρχει ένα σημείο το οποίο μου φαίνεται ιδιαίτερο θα έλεγα αδύναμο στη, στα πρακτικά μέτρα τα οποία προτείνεται και αφορά το περιβάλλον. Υπάρχουν κάποιες περιφέρειες οι οποίες έχουν δικά τους περιβαλλοντικά προγράμματα, οι οποίες ενεγράφησαν στα πλαίσια της ε, λογικής της Κοπενχάγης και αυτό πρέπει να είναι μια προτεραιότητα και για την αναδιάταξη την οποία εσείς προτείνετε, γιατί δεν τα συμπεριλαμβάνετε αυτά τα μέτρα. Πέραν της προσπάθειας που έκαναν και τα κράτη-μέλη με τα οποία συνεργαστήκατε για να εξεταστεί συνολικά η κατάσταση, θα θέλαμε να υπάρξει μια διαβούλευση και με τις περιφέρειες, γιατί θυμίζω ότι σε επίπεδο περιφερειακό εκτελούνται τα προγράμματα. Vážený komisaři, paní předsedkyně, dovolte, Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ καλή η ευκαιρία που έχουμε να συζητήσουμε μαζί σας τα θέματα αυτά. Να σας θέσω μια ερώτηση κύριε Επίτροπε. Είπατε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσει κανείς να απλουστεύσει τους κανόνες, ιδιαίτερα σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και τους διαγωνισμούς τους κρατικούς, εκεί όπου δημιουργούνται και τα περισσότερα προβλήματα και οι περισσότερες τρευλώσεις. Έχετε καταλήξει σε μια κατάσταση των πραγμάτων σε σχέση με τον τρόπο που διεξάγονται οι διαδικασίες αυτές εσείς πιστεύετε ότι τα κράτη-μέλη είναι σε θέση ή είναι ήδη στη διαδικασία απλούστευσης των διαδικασιών ή μήπω η προσπάθεια η οποία γίνεται έχει παραμείνει σε επίπεδο Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Τώρα για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση. Η διαδικασία που προτείνατε πράγματι είναι κάτι που βελτιώνει τον τρόπο χρήσης των Ευρωπαϊκών Ταμείων και γι' αυτό θέτω εδώ την ερώτηση. Στο μέλλον, πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε περαιτέρω εγγυήσει για την εφαρμογή των αρχών που ακολουθήσαμε μέχρι τώρα στην πολιτική συνοχή. Μια τρίτη ερώτηση αφορά την εναρμόνιση των κανόνων για τη χρήση των μεμονωμένων ταμείων. Παράδειγμα για να με καταλάβετε. Η χρήση πόρων που προέρχεται από τον αγροτικό τομέα. Εκεί δεν υπολογίζεται το ΦΠΑ σαν παράδειγμα ενώ ακριβώς το ΦΠΑ σε άλλα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από άλλα ταμεία υπολογίζεται το ΦΠΑ. Αυτές λοιπόν οι διαφορές πώς θα αντιμετωπιστούν στο μέλλον. Και μια τελευταία ερώτηση. Το θέμα της ευελιξίας είναι προς στιγμή ένα θέμα που αντιμετωπίζεται σαν αρχή, σαν θεωρία. Πρακτικά, τι θα κάνετε με αυτό στο μέλλον. Νομίζω ότι ο επόμενος που έχει δει στο λόγο είναι Απόν. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. And uh, Μπάφτον, για την ενδιάμεση αναθεώρηση. Έχω κάποιες ανησυχίες μεσοπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες. Κύριε Χάν, μας εξηγήσατε ότι υπάρχουν κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούνται και τα οποία αφορούν τις δυνατότητες ε, που έχουν τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν στις χρηματοδοτήσεις. Ε, φοβόμαστε ότι δεν θα υπάρχουν ε, τα χρήματα αυτά, τουλάχιστον σε ορισμένες χώρες, και αναφέρομαι στη δική μου συγκεκριμένα. Εσείς τους μήνες που είσαστε στη θέση σας έχετε δει κάτι το οποίο να σας καθησυχάζει προς την κατεύθυνση αυτή μπορείτε να μας δώσετε τη δική σας ερμηνεία για τις δυνατότητες ε, της χρηματοδότησης από την πλευρά των κρατών, κ. Σταυρακάκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι λακωνικότατος. Έχω δύο ερωτήσεις. Κύριε Επίτροπε, πιστεύετε ότι το δικό σας όρομα για το μέλλον της πολιτικής συνοχής που μας παρουσιάσατε θα τεθεί σε περίοπτη θέση στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές. Σε ό,τι αφορά το μερίδιο που θα έχει στον προϋπολογισμό αυτή η πολιτική συνοχής. Δεύτερη ερώτηση. Σημαντική είναι η πολιτική συνοχή, αλλά πολύ σημαντική είναι και εξασφάλιση τη ενεργειακή μα ανεξαρτησία και η υλοποίηση των στόχων του 2020 για τι κλιματικέ αλλαγέ στην δημοσιονομική αναθεώρηση, πού θα βρείτε τα συμπληρωματικά κονδύλια ε, στον προϋπολογισμό για την ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές. Μπορεί, πιστεύετε ότι μπορεί ο προϋπολογισμός να φτάσει στο 1,24 του ΑΕΠ, να ξεπεράσει λίγο το ανώτατο όριο που έχουμε συμφωνήσει θα πρέπει να γίνουν περικοπές στις ε, υπάρχουσες πολιτικές. Και αν ε, θα γίνουν περικοπές, από ποιες πολιτικές θα γίνουν αυτές οι μειώσεις των δαπανών. Ευχαριστώ κύριο Επίτροπος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αλφόνζη, καταρχήν να απαντήσω σε εσά. Για παράδειγμα, ε, πέρσι 80 επιχειρησιακά προγράμματα αναπροσαρμόστηκαν με βάση τις ανάγκες που εντοπίστηκαν στις διάφορες περιφέρειες. Τα επιχειρησιακά προγράμματα μετά την υιοθέτησή τους δεν σημαίνει ότι είναι πλέον κλειδωμένα αν θέλετε. Δηλαδή εάν υπάρχει κάποια ανάγκη διόρθωσης, η διόρθωση αυτή λαμβάνει η χώρα χωρίς βέβαια να θέλουμε και επενθυμίζουμε πάντοτε να μην χάνεται η διάσταση της στρατηγικής μέσα από μια τέτοια διορθώση. Σε ό,τι αφορά τα έργα στον χώρο της περιβαλλοντικής ε, πολιτικής ε, δεν ε, οφείλεται κάτι τέτοιο κατά πρώτο λόγο στην περιφερειακή πολιτική την ίδια αλλά στις εθνικές νομοθεσίες για το περιβάλλον οι οποίες συχνά δεν συνάδουν με ε, τις ε, κοινωτικές διατάξεις και κατά συνέπεια δεν υπάρχει η, βάση, η νομική βάση για την αξιοποίηση κοινωτικών ε, κοντιλίων. Άρα λοιπόν αυτό που θα πρέπει να διασφαλίσουμε είναι ότι να μην χρειάζεται, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τα νέα να γίνονται τέτοιες αναπροσαρμογές νομοθετικές. Ο ε, συνάδελφος ε, κύριος ε, Ποτότσινεκ είχε απευθυνθεί μάλιστα σε μένα, μου είχε θέσει μια σχετική ερώτηση και έχουν δοθεί σχετικέ εντολέ στου δύο γενικού διευθυντέ, ούτω ώστε να αναζητηθεί εδώ ένα κοινό παρανομαστή για τη συνεργασία. Εάν και εδώ μεθαίνουν στον κύριο Σταυρακάκη και εφόσον αυτά τα προγράμματα αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του συνολικού μας προπολογισμού, αυτά δηλαδή για το περιβάλλον. Τώρα, σε ό,τι αφορά το public procurement θα πρέπει να γίνει ε, μια αποκοινού εξέταση με την Γενική Διεύθυνση Μάρκ ως προς το ε, τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε. Ήδη έχουμε προβεί κάποια βήματα σε ό,τι αφορά δηλαδή τις ε, απλουστεύσεις ε, ειδικότερα σε ό,τι αφορά ε, έργα με μικρότερο προϋπολογισμό και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο τα μέτρα αυτά λειτουργούν και αξιοποιούνται ε, μια σχετική δήλωση από την δική μου πλευρά είναι λίγο πρόωρη αυτή τη στιγμή, δηλαδή με βάση το, τα έγγραφα που λαμβάνουμε θεωρούμε πως λειτουργούν γιατί αλλιώς δεν θα γινόταν αυτές οι προτάσεις αλλά ε, ξέρετε δεν είναι πάντοτε έτσι δεν θέλουμε δηλαδή με αυτήν την απλούστευση να οπισθοδρομήσουμε και να γυρίσουμε σε προηγούμενες ε, πρακτικές άρα χρειάζεται εδώ μια ισόρροπη προσέγγιση σε ό,τι αφορά τώρα το integrated approach αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση προσπάθησα να ανταποκριθώ σε αυτό καλώντας από νωρίς τους συναδέλφους επιτρόπους και τις γενικές τους ε, όχι μόνο κατά την εκπόνηση του προγράμματος εργασιών αλλά και στη φάση της υλοποίησης και του monitoring, της παρακολούθησης ούτως ώστε οι στόχοι τους οποίους έχουμε θέσει και οι προτεραιότητες που έχουμε θέσει να εφαρμόζονται με ευελιξία στις ε, περιφέρειες αλλά ταυτόχρονα και να διατηρούνται γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό ε, να έχουμε κατανοήσει νου Έχουμε ήδη μια καλή εδώ απόδοση performance, αλλά θα πρέπει τώρα να περάσουμε στο, στην αισίαση στο αποτέλεσμα, δηλαδή του να εξετάζουμε το κατά πόσο τα, οι στρατηγικοί στόχοι ε, υλοποιούνται μέσω των επιμέρους ε, προγραμμάτων και αυτό απαιτεί την συνεργασία μέχρι ενός σημείου και των υπολείπων γενικών διευθύνσεων. και εδώ ε, η στάση των άλλων επιτρόπων και των οικών διευθυνσεών ε, και η πρόθεσή τους να ε, έχουμε εδώ μια τέτοια συνεργασία είναι πολύ θετική και ελπίζω πως σωματικά αυτή η πρακτική, αυτή η προσέγγιση θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Και εδώ ε, εδώ έχουμε και το ζήτημα της συνεργασίας του ανθρώπου σε ό,τι αφορά τον ε, χώρο της αγροτικής ανάπτυξης ε, και τους άξονες 3 και 4, τους περιβόητους, ώστε να οδηγηθούμε εδώ σε ένα καλύτερο συντονισμό μεταξύ μας. Μπορούμε να μιλήσουμε ενδεχομένω εδώ και μια ένα ρόλο ηγετικό τον οποίο θα αναλαμβάνει η κάθε πλευρά σε ό,τι αφορά επιμέρους ζητήματα. Αλλά από εκεί και μετά εγώ δεν θέλω να ε, επενδύσω εδώ ε, τις δυνάμεις μου στην κατανομή αν θέλετε αρμοδιοτήτων θέλω να επενδύσουμε καλύτερα στην ίδια ουσία. Σε ό,τι αφορά την ενδιάμεση αναθεώρηση, ήδη αναφέρθηκα ότι ναι, εμείς έχουμε εδώ ένα σημαντικό ρόλο. Ε, κύριε Μπάφτον, ε, δεν αντιλαμβάνομαι αυτό που ρωτήσατε, ότι δηλαδή για την Ιουαλέα δεν υπάρχουν τα κατάλληλα κοντήλια Το ερώτημα είναι το κατά πόσο η Ιουαλέα είναι στη θέση να δεσμεύσει αυτά τα κοντήλια για ε, γενικά πάντως η περιφέρεια αυτή η δηλαδή δεν μας δημιουργεί προβλήματα. Τώρα σε ό,τι αφορά την ενέργεια και την διασφάλιση της ενεργειακής μας αυτονομίας και τον μελλοντικό προπολογισμό ε, δεν νομίζω να εκπλαγείτε να σας πω ότι δεν μπορώ να σας πω κάτι αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ο Επίτροπος από τον προπολογισμό μπορεί να σας πει κάτι σε αυτή τη φάση. Προφανώ ότι εδώ προσπαθούμε να διασφαλίσουμε περισσότερα κονδύλια. Είναι αυτονόητο, αλλά και σε αυτόν τον τομέα υπάρχει μια καλή συνεργασία στην ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί έχουμε κοινού στόχου. Και ο τρόπος της υλοποίησης είναι σημαντικός, αποτελεί κάτι το πρωταρχικό, γιατί σχετίζεται με τη βιωσιμότητα. Δηλαδή, ναι, με ένα αναθεώρηση του περιεχομένου, αλλά στο πλαίσιο μια κοινή προσέγγιση, ενό integrated approach, γιατί ε, μόνο με αυτόν τον τρόπο ε, μπορούμε να υλοποιήσουμε του συνολικού μα στόχου. ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Χισμένοβα, φίλη Κύριε Επίτροπε, ποια είναι η γνώμη σας για την πολιτική συνοχή μετά το 2013, σε ό,τι αφορά τις φτωχότερες περιφέρειες της Ένωσης. Και ποια είναι τα μέσα, τα εργαλεία και, του, και τους μηχανισμούς που θα χρησιμοποιήσουμε για να καταπολεμήσουμε αυτήν την υστέρηση ορισμένων περιοχών και τις ανισότητες. Η κυρία Ελίζα Βεσρέντερ και μετά ο κύριος Μιχάλης Τρεμόπουλος. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Τρία σύντομα ερωτήματα. Πρώτο, κάτι το οποίο αφορά αυτό στο οποίο ήδη αναφερθήκατε. Δηλαδή μεγάλα έργα και νομοθεσία περιβαλλοντική. Μα είπατε πω υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν ακόμα μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο ορισμένε ε, κοινωτικές διατάξει για το περιβαλλον. Ε, δηλαδή τι σημαίνει σε αυτή την περίπτωση, δεν ισχύουν, δεν εφαρμόζονται για τα μεγάλα έργα και σε αυτή την περίπτωση α, υλοποιούνται κανονικά, εγκρίνονται. Ε, δεύτερον, σε ό,τι αφορά τη στατική έκθεση, εκεί λοιπόν αναφέρεται στην έκθεση ότι σε πολλές εκθέσεις και σε πολλές συζητήσεις αναφέρεται αυτό το ζήτημα της εταιρική σχέσης. Υπάρχουν δηλαδή και κάποιες εκθέσεις και κάποιες συζητήσεις στις οποίες δεν συζητείται, δεν θίγεται κάτι τέτοιο. Τρίτο ερώτημα και πάλι στη στρατηγική έκθεση. Αναφερθήκατε στο ποσοστό των γενικών στο MSF αλλά όχι στο ΕΦΡΕ. E. Γιατί ε, θα θέλαμε να, να μας πείτε εδώ, να μας δώσετε ε, περισσότερες πληροφορίες, δηλαδή τι μας λέτε σε αφορά τις ε, σχέσεις απέναντι σε γυναίκες συγκεκριμένα. Ο κύριο Μιχάλη Τρεμόπουλο και μετά Λούχαν. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα εστιάσω σε ορισμένου τομεί τη περιφερειακή πολιτική με στοιχεία συγκεκριμένα από την στρατηγική αναφορά του 2010 τη Κομισιόν για την Πολιτική συνοχή Στον τομέα τη ενέργεια και στο θέμα της ε, Community Strategic Guidelines ε, το επίπεδο της προόδου βλέπουμε ότι είναι ιδιαίτερα χαμηλό και πολλά κράτη-μέλη βρίσκονται σε κατάσταση σημαντικών ε, καθυστερήσεων με μικρή και καθόλου πρόοδο. Μεταξύ αυτών και η χώρα μου, η Ελλάδα. Το, επίσης, το συνολικό ύψος των επενδύσεων στο περιβάλλον υστερεί. Ο όγκος των σχεδίων που έχουν επιλεγεί ε, στο θέμα της ε, Community Strategic Guidelines ε, φτάνει το 21% και ορισμένα κράτη-μέλη, μεταξύ τους πάλι και η Ελλάδα, αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των σχεδίων. Σε επίπεδο κλάδου, ενώ οι επενδύσεις στην επεξεργασία των λιμάτων αποδίδουν 27,5% έχουν διατεθεί εκτός από κάποιες χώρες, μεταξύ τους και η Ελλάδα με 5,5, στο στάδιο πρόληψης του κινδύνου και αποκατάστασης των βιομηχανικών χώρων και των μολυσμένων εκτάσεων, υστερούν και πάλι. Στον τομέα αυτό, σε κάποιες χώρες, την πρόληψη κινδύνου, σε κάποιες χώρες λοιπόν είναι ιδιαίτερα ασθενής η απορρόφωση μεταξύ τους, μεταξύ τους πάλι και η Ελλάδα. Και τέλος, η πρόοδος όσον αφορά την επιλογή των ε, σχεδίων για τις πολιτιστικές και κοινωνικές υποδομές, δηλαδή τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τα κοινωνικά κέντρα, ε, έξι χώρες αναφέρουν πρόοδο άνω του μέσου όρου και, κάποια, και οι άλλες πέντε έχουν μείνει πολύ πίσω. Μεταξύ τους πάλι η Ελλάδα. Ρωτώ, πού οφείλεται αυτή η στέρηση. Μπορεί να θεραπευτεί. Και τι προτίθεστε να κάνετε ώστε να υπάρξει κάποια πρόοδος. Ο και μετά η Ερικα ε, Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για τα συγκεκριμένα ε, στοιχεία που μας δώσατε τώρα σε ό,τι αφορά τα νέα χρηματοδοτικά μοντέλα μας αναφερθήκατε στις νέες ευκαιρίες που μας δίνονται και στην ε, κατανομή των ε, κονδυλίων, ε, πράγμα το οποίο είναι πολύ θετικό γιατί γνωρίζουμε ότι πράγματι κάθε περιφέρεια έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και γι' αυτό θεωρούμε πως ε, θα ήταν η καλύτερη δυνατή λύση να έχουμε αντίστοιχα κονδύλια, αντίστοιχη κατανομή, ώστε να επιτυχάνουμε μεγαλύτερη, καλύτερη απόδοση. Η δική μου ερώτηση είναι υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο μία τέτοια λίστα, αν θέλετε, ανακών και από εκεί και μετά μια λίστα με ε, ιεράρχηση προτεραιότητας ε, των διαφόρων αναγκών των περιφερειών και των κρατών μελών. Και αν υπάρχει μια τέτοια λίστα, οι σχετικές χρηματοδοτήσεις έχουν ή θα προσανατολιστούν με βάση αυτές τη σημασία των διαφορετικών αναγκών και αν δεν το έχετε κάνει ακόμα πότε θα το κάνετε. Η κυρία Ρίκα Μάνερ. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για την εμπεριστατωμένη παρουσίαση και τις πολύ μεστές απαντήσεις που δώσατε. Αναφερθήκατε στις μακροπεριφέρειες. Θα ήθελα να μας δώσετε περισσότερες εξηγήσεις. Ποιο είναι το μακροπρόθεσμο σε σχέδιο και όραμα για αυτές τις μακροπεριφέρειες και ποια είναι η σχέση των μακροπεριφερειών με τα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης. Για παράδειγμα, έχουμε ήδη τέτοιο πρόγραμμα για τη Βαλτική θάλασσα. Μπορείτε να αναφερθείτε λίγο και στη χρηματοδότηση. Επαναλαμβάνω, ποιε είναι οι προθέσει μακροπρόθεσμα για τι μακροπεριφέρειες και πώ θα συνδέσετε και θα συνδυάσετε τι διάφορε πολιτικέ. Για τι μακροπεριφέρειες και πάλι και για τη Βαλτική. Γνωρίζετε ότι εκεί εφαρμόζεται ένα πολύ σημαντικό πιλωτικό πρόγραμμα για μακροπεριφέρεια πολύ μεγάλο επίβολο πρόγραμμα και φαντάζομαι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθήσει εκ του στην εφαρμογή του. Ευελπιστώ ότι και εσείς θα συντάξετε ένα έγγραφο με σχολιασμό αυτής της εφαρμογής, γιατί προς το παρόν δεν υπάρχει τίποτα. Σκοπεύετε να δημοσιεύσετε ένα σχετικό έγγραφο για το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα της Βαλτικής. Γνωρίζετε το άρθρο 74 της Συνθήκης της Λισαβόνας, που αναφέρεται στην περιφερειακή πολιτική που θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των ευρωπαϊκών περιφερειών και των πιο απόμακρων και φτωχών. Θα είναι όντως ε, πανευρωπαϊκό αυτό αυτή η προσέγγιση, πανευρωπαϊκή προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Περιφέρειες. Ja, zum Thema Kohäsion. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ε, πολιτικής ε, συνοχής ε, μετά το 2013, επανειλημμένα έχω αναφερθεί σε αυτό. Η λόγο πολιτική θα πρέπει να συνεχιστεί και δεν είμαι ιδιαίτερα ευτυχή με το γεγονό ότι κάνουμε συνέχεια λόγο για προγραμματικέ περιόδου. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε κατά νου μια συνεχή ε, πολιτική στο πλαίσιο βέβαια της οποίας ε, λαμβάνει η χώρα ένας έλεγχος ή μια αναθεώρηση, αναπροσαρμογή ε, των διαφόρων στοιχείων και της καλής λειτουργίας ή όχι. Αλλά η ερώτηση που τίθεται ανατακτά χρονικά διαστήματα σε ό,τι αφορά τον πυρήνα της ειδικής πολιτικής νομίζω πως είναι περιττή. Η περιφερειακή πολιτική αποτελεί κατά κύριο λόγο μια αρχή πολιτικής ε, την οποία καλούμαστε να εφαρμόζουμε ξανά και ξανά. Δεν πρόκειται λοιπόν για κάτι το οποίο ισχύει ε, μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία και από εκεί και μετά ε, θεωρείται πως έχει περατωθεί, έχει ολοκληρωθεί, έχει επιτύχει. Πρόκειται για μια αρχή σε ό,τι αφορά την πολιτική, η οποία θα πρέπει να έχει μια συνεχή ισχύ, καθώς αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της ευρωπαϊκής πολιτικής της χαράξης της. Άρα ε, θα ήθελα να βρούμε μια δυνατότητα να ξεφύγουμε λίγο από αυτήν την εκθεμελίων, αν θέλετε, επανεξέταση της ειδικής πολιτικής ανά 7 χρόνια και καλύτερα να κινηθούμε προς μια συνεχή πολιτική. Σε ό,τι αφορά τώρα τα μεγάλα έργα, γι' αυτό αναφέρθηκα σε αυτά. Εάν δεν υπάρχει ε, ευθυγράμμιση με την ε, εθνική και κοινωνική πολιτική, δεν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης. Ε, και η Γενική Διεύθυνση ε, Περιβάλλοντος ξέρει τι θα πρέπει να συμβεί εκεί. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν οι εθνικές προϋποθέσεις για εφαρμογή τέτοιων ε, έργων. Αλλά θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν κάποιε μεταβατικέ περίοδοι, οι οποίε είναι ακριβώ αυτό, μεταβατικέ. Δηλαδή, μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πρέπει να υπάρχει εφαρμογή ε, παρόλα αυτά όμω σα λέω σε ορισμένε περιπτώσεις δεν έχει λάβει χώρα αυτή η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, αυτή η υλοποίηση και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η υλοποίηση και των αντίστοιχων έργων. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, την συμμετοχή γυναικών στο ΕΦΡΕ, από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχουν κάποια στοιχεία ε, από όσο γνωρίζω σας λέω γιατί κυρίως εδώ οι ενισχύσεις κατευθύνονται προς φορείς ενώ στο MDF έχουμε ας πούμε, περισσότερα, το μεγαλύτερο μέρο των κονδυλίων να κατευθύνεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα, ούτως ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει σε ό,τι αφορά δηλαδή, την κατανομή. Ε, σε ό,τι αφορά ε, ε την Ελλάδα συνολικά. προφανώ αντιλαμβανόμαστε ε, την, ε, ότι η κρίση εδώ παίζει ένα σημαντικό ρόλο και στο επίπεδο της χρηματοδότησης ως προς το κατά πόσο δηλαδή είναι δυνατή η χρηματοδότηση και η υλοποίηση έργων ή όχι. Αλλά εάν ε, δημοσιεύουμε καταλόγους με ε, κράτη-μέλη, προφανώς κάποια θα βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο και κάποια κάτω από το μέσο όρο. Δηλαδή είναι πολύ ασυνήθιστο το να βρίσκονται όλοι κάπου ε, στο μέσο όρο. Ε, προσπαθούμε δηλαδή αν θέλετε να παράσχουμε τα κίνητρα εκείνα που χρειάζονται για εκείνους οι οποίοι κατά τη φάση της δημοσίευσης μιας έκθεσης βρίσκονται κάτω από το μέσο όρο. Ε, με αυτόν τον τρόπο δηλαδή ε, ε συνεισφέρουμε, ε, ταρακουνάμε δηλαδή λίγο όσους βρίσκονται κάτω από το μέσο όρο, αλλά προσπαθούμε και σε ό,τι αφορά τι επιχειρησιακέ ε, λεπτομέρειε και στο επίπεδο του capacity building, τη δημιουργία δηλαδή των αντίστοιχων δυνατοτήτων και υποδομών, γιατί σίγουρα και αυτό αποτελεί πρόβλημα, πέρα από την ε, χρηματοδοτική κατάσταση να συμβάλλουμε. Αλλά προφανώ η οικονομική κατάσταση, αυτή η διάσταση είναι πολύ σημαντική σε αυτή τη φάση για την Ελλάδα, αλλά και γι' αυτό είπα και εγώ από την δική μου πλευρά πως εμ, τα ε, κονδύλια από τα διαφθορτικά ε, ταμεία δεν ε, θα έπρεπε να αποτελέσουν το, το κύριο σημείο που δίνεται έμφαση. Θα πρέπει να συνεχίζεται κανονικά να υπάρχει η χρηματοδότηση και η υλοποίηση των σχετικών έργων ώστε να συμβάλλουν αυτά τα κονδύλια στην ανάκαμψη. Σε ό,τι αφορά τα απαραίτητα τώρα κονδύλια δεν έχουμε ακόμα αναλογιστεί κατά πόσο δηλαδή το ένα κράτος μέλος ή το άλλο ε, κράτος μέλος ε, χρειάζεται τα τάδε τα δίνα κονδύλια. Προσπαθούμε να έχουμε ε, διαθέσιμα συνολικά τα απαραίτητα κονδύλια και μέσα στην τελευταία περίοδο υπήρξε δεκαπλασιασμός του σχετικού εργαλείου Αλλά για να ξέρουμε γιατί μιλάμε εδώ, γιατί νούμερα μιλάμε ότι πήγε από το 1 δισεκατομμύριο στα περίπου 11 δισεκατομμύρια στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Άρα λοιπόν σημαντική αύξηση, αλλά ε, σε ό,τι αφορά το, το ύψος ως ποσοστό του προπολογισμού παραμένει μικρό. και ίσω στο πλαίσιο του Financial Engineering και τη ίδια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γίνεται αντιληπτό λίγο με διαφορετικό τρόπο αυτό το, το, το εργαλείο αν θέλετε σε σχέση με κάποιου άλλου που έρχονται από το χώρο τη ιδιωτική οικονομία. Εν πάση περιπτώσει το Financial Engineering ε, κατευθύνεται ακριβώς στην δημιουργία τέτοιων εργαλείων τα οποία συνάδουν με την ε, κοινωτική νομοθεσία και τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν, μπορούν να αξιοποιηθούν και να υλοποιηθούν από την πλευρά των κρατών μελών. Δεν είναι πρόθεσή μας δηλαδή να λέμε στο α κράτο μέλος χρησιμοποιήστε αυτό ή εκείνο το εργαλείο ενώ το άλλο το, το β κράτο μέλος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει διαφορετικά εργαλεία. Εκείνο το οποίο εμεί θα κάνουμε είναι να δίνουμε συστάσει ω προ το ποια εργαλεία του financial engineering είναι κατάλληλα για ποιο είδο έργων. έργων συγγνώμη για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την κατασκευή πανεπιστημίων. Δεν πρόκειται για κάτι, για ένα είδος ε, προγράμματος το οποίο θα πρέπει να σκεφτούμε την αναχρηματοδότηση. Αλλά σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την κατασκευή ενός αυτοκινητόδρομου, προφανώς μέσω ε, τελών, μέσω διότι να αναλογιστούμε το ενδεχόμενο της αναχρηματοδότησης. Άρα λοιπόν η προσπάθεια που γίνεται είναι μεταξύ άλλων ποια είναι τα ίδια γίνει έργα τα οποία θα πρέπει να έχουν και αυτό το στοιχείο της αναχρηματοδότησης περισσότερα, περισσότερους τρόπους financial engineering. Εκείνο όμως που θα πρέπει να δούμε ε, είναι το πώς μπορεί να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα το, το, το μοντέλο της ε, ιδιωτικής δημόσιας εταιρικής σχέσης του public-private ε, ε, partnership. Νομίζω πως ε, αυτό το μοντέλο έχει, δεν έχει ενισχυθεί τόσο πολύ. Έχει υποχωρήσει λίγο και θεωρώ αυτό που συμβαίνει επειδή επειδή οι επιχειρήσεις οι οποίες βλέπουν ότι για την χρηματοδότηση ενός συγκεκριμένου έργου υπάρχει ένα βάθος χρόνου 30 ετών δημιουργεί δυσκολίες για τους ίδιους τους επιχειρηματίες, δημιουργεί μια ανασφάλεια δηλαδή. Πρόκειται για ζητήματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε στην Σε ό,τι αφορά τώρα τις μακροπεριφέρειες, είπαμε πως έχουν ε, κάποιες ε, πρωτοβουλίες οι οποίες ξεκίνησαν σε συγκεκριμένες περιφέρειες και αυτό λοιπόν σημαίνει ότι δεν έχουμε τον ε, σκοπό εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρουμε το χάρτη της Ευρώπης και να πούμε να μια μακροπεριφέρεια που θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ή να μια άλλη. γιατί ε, αν δούμε κοινά ενδιαφέροντα αν θέλετε περιφερειών προφανώς θα μπορούσαμε να έχουμε μεγάλο αριθμό ε, διαφορετικών μακροπεριφερειών τις οποίες θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε αλλά αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε πώς λειτουργούν τα πράγματα και σε ό,τι αφορά τη στρατηγική ε, για την Βαλτική μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2011 θα υπάρξει μια σχετική έκθεση η οποία θα εξετάσει ακριβώς αυτό, δηλαδή το πώς έχουν ελοποιηθεί τα σχετικά έργα και το ποια είναι η αναμένω πως θα είναι η βιωσιμότητά τους. Νομίζω πως απάντησα σε όλα τα ερωτήματα. Ευχαριστώ Επίτροπε. Άλλοι 13 έχουν ζητήσει το λόγο και δεν έχουμε πάνω από 10 λεπτά για όλους σας. Εσείς προσπαθήστε να, είναι σύντομος, να είστε σύντομος, το αναγνωρίζω. Εν πάση περιπτώσει, όχι πάνω από μισό λεπτό για την ερώτησή σας, όχι σχόλια, γιατί αλλιώς θα καθυστερήσουμε να περάσουμε στο επόμενο επίσης σημαντικό θέμα. Και πριν το καλοκαίρι ο Επίτροπος θα επανέλθει στην Επιτροπή μας, ως εκ τούτου θα έχουμε δυνατότητα περαιτέρω συζητήσεων. Λοιπόν, συντομέσετε παρακαλώ τις ερωτήσεις σας από εδώ και πέρα. Ja, Vorsitzende, sehr geehrter Kommissar, vielen Dank Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ε, καταρχήν σα ευχαριστούμε για το ότι έχετε καταστήσει αντικείμενο δύο εκθέσεων και το ζήτημα τη καινοτομία. Δύο ερωτήματα. Σε ό,τι αφορά την έγκριση ε, κονδυλίων και τη ροή των κονδυλίων από την πλευρά του ΕΦΡΕ, Βλέπουμε ότι υπάρχουν εδώ μια, πια μια θετική εξέλιξη, αλλά έχουν ε, αναφερθεί και κάποιες δυσκολίες. Ε, θα μπορούσατε να μα πείτε σε ποιε περιφέρειες ε, έχουν εντοπιστεί αυτέ οι δυσκολίε. Θα μπορούσατε να μας διαθέσετε τουλάχιστον αυτές τις πληροφορίες. Και μετά, σε ό,τι αφορά την ε, προηγούμενη περίοδο, όπου έγιναν κάποιε επικριτικέ ε, παρατηρήσει από την πλευρά του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα θέλαμε να ξέρουμε τι έχει συμβεί. Και δεύτερη ερώτηση, ε, σε ό,τι αφορά την έκθεση Άρκα, ποια είναι η δική σα θέση, τι νομίζετε πώ θα συμβεί από εδώ και πέρα. Ο Φράνσο το λόγο, μισό λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστούμε την Επίτροπα ΕΧΑΝ για τις ε, σαφείς τοποθετήσεις σας. Θα ήθελα να θέσω ένα ζήτημα εδώ και ένα ερώτημα. Οι συνάδελφοι από τη στρατηγική για τον Τούναβη να μας ε, διαθέσουν αν θέλετε τις πληροφορίες σε ό,τι αφορά τα σχετικά έργα που έχουν ολοποιηθεί από κοινού σε μια κοινή ανακοίνωση. Νομίζω πως κάτι τέτοιο θα ήταν ε, πολύ χρήσιμο και για τη διάσκεψη, δηλαδή να έχουμε μια συνολική παρουσίαση αυτών των έργων. Ε, το ερώτημά μου τώρα. Ε, ήδη το αναφερθήκατε σε αυτό, αλλά θα ήθελα να λάβω μια διευκρίνηση σε ό,τι αφορά τις, ε, τις ε, περικοπές σε ό,τι αφορά τις ε, ενισχύσεις σε περιφέρειες, σε ό,τι αφορά κάποιους οι οποίοι έχουν προβεί σε παραβάσεις, ε, ε, ποια θα είναι η δική σας θέση. Μας είπατε πως δεν θα υπάρξουν κανένα είδους περικοπές για διάφορες περιφέρειες, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Είπατε πως θα πρέπει να, συνεχιστεί, να συνεχιστούν οι επενδύσεις και θα πρέπει να υπάρχουν και θα πρέπει να έχουν ισχύσει αυτό το μοντέλο. Αλλά ε, ε, πώς να αντιληφθούμε τα όσα είπε ο κύριος Ερέν ε, στις 14 Απριλίου, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει ενδεχομένως θα πρέπει να λογιστούμε και κάποιες περικοπές σε ό,τι αφορά συγκεκριμένες περιφέρειες οι οποίες έχουν κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά τον Το λόγο έχει ο κύριος παρακαλώ. Χρόνο φίδο. τρία ερωτήματα, πει. Ε, τι θα κάνει ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά ε, τα 30 επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία δεν έχουν ακόμα εκδοθεί και τα οποία αφορούν συγκεκριμένα κράτη-μέλη, τα οποία είναι δηλαδή αφορούν συγκεκριμένε εδαφικέ επικράτειε, δεν είναι διασυνοριακά. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Δεύτερο, ε, εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή εν Ε, και η, ε, το δικό μας ποσοστό απορρόφησης ε, βρίσκεται στο 25 με 30%. Ε, μας λέτε ότι έχουν γίνει ήδη κάποιες προκαταβολές, αλλά εάν σας λέω ο ρυθμός της απορρόφησης παραμένει τόσο χαμηλός, τι ακριβώς θα κάνετε. Ε, και μετά σε ό,τι αφορά την έκθεση θα δώσετε κάποια συνέχεια σε αυτήν την ε, περιφέρεια, ε, συγγνώμη, σε αυτήν την έκθεση. Δεν μας το διευκρινίσατε αυτό. Ευχαριστώ. Βόιτσο Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, είπατε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει σε μεγαλύτερο βαθμό να υλοποιήσουν τους στόχους πολιτικής συνοχής και απευθύνεται έκκληση προς τα κράτη-μέλη. Αυτό προσπαθούν φαντάζομαι, αλλά τι βαθμό δέσμευση υπάρχει από τα, από τα επιμέρους ό,τι αφορά την υλοποίηση των στόχων τη πολιτική συνοχή και τη περιφερειακή πολιτική. Και δεν μιλώ μόνο για τα κοινοτικά κονδύλια, τα κονδύλια από τον κοινοτικό προπολογισμό, αλλά τι επιπλέον δεσμεύσει από του εθνικού προπολογισμού. Γιατί αν παρακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία θα μπορέσουμε να συγκρίνουμε και τις δυσαναλογίες που υπάρχουν στην πολιτική, περιφερειακή πολιτική και στην πολιτική συνοχή. Γιατί στην Πολωνία, για παράδειγμα, και για τις δύο πολιτικέ ε, επαφιόμαστε στην ε, Ένωση κυρίω, στα κοινωτικά κονδύλια. Ενώ φαντάζομαι για την πολιτική του 2020 ε, προϋποθέτει μια τέτοια ανάμειξη μεγαλύτερη από τον εθνικό προϋπολογισμό. Αλλά στο μέτρο που δεν δεσμεύονται εξίσου όλα τα κράτη-μέλη θα επιταθούν οι ανισότητες και τις αναλογίες μεταξύ των διαφόρων χωρών μελών. Ο κύριο Γιάννα Αλμπρίχτ. Έχω τρει ερωτήσει, κύριε Επίτροπε. Και μία σύσταση. Παρόλο που είπατε ότι δεν θα πρέπει να εκφέρουμε όψη γιατί δεν προλαβαίνουμε. Πρώτη ερώτηση. Ό,τι αφορά την υλοποίηση τη πολιτική ε, για την περίοδο 2007-2013. Κύριε Επίτροπε, πιστεύετε ότι θα πρέπει στην περίοδο αυτή να γίνουν κάποιες αλλαγές στα συστήματα εφαρμογής, στη διάρκεια της περίοδου προγραμματισμού. Ακόμη και πριν το 2013 θα πρέπει να αλλάξει το σύστημα. Δεύτερη ερώτηση. Τι γίνεται με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ο αρμόδιος επίτροπος πιστεύει ότι το Κοινωνικό Ταμείο θα πρέπει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής. Τρίτη ερώτηση. Στην πέμπτη έκθεση Μπορούμε να περιμένουμε, όπως και στην τρίτη έκθεση, να περιληφθεί πρόταση συστημική για το 2013 ή θα γίνουν μόνο κάποιες ε, εισαγωγικές παρατηρήσεις. Και η σύστασή μου είναι ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη το συντομότερο δυνατόν και με πολύ κατηγορηματικό τρόπο να διαλευκανθεί το θέμα της στρατηγικής για τη Βαλτική και το Δούναβι, γιατί ακροθυγώς μόνο το αναφέρεται. Εγείρονται ελπίδες και προσδοκίες ε, για χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων. Θα πρέπει όμως να είμαστε σαφείς και κατηγορηματικοί, γιατί έχουμε μια, είχαμε, έχουμε μια πραγματικά νέα ευρωπαϊκή στρατηγική και έχουμε πραγματικά προγράμματα στα πρέσια του τρίτου στόχου ο κύριος Μποστινάρου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, πολιτική συνοχής, ε, συνδεσιμότητα, κινητικότητα. Και την περασμένη εβδομάδα όμως είχαμε το ηφαιστιακό, νέφος, ε, το, το νέφος με τις ηφαιστειακές ε, στάχτες που μας αναστάτωσε όλους. Επίσης έχουμε αντίστοιχα προγράμματα, τεράστια αναπτυξιακά προγράμματα στην Κίνα ή στις Ηνωμένε Πολιτείες Πιστεύετε ότι στις, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουμε στο μέλλον τέτοια μεγάλα επίβολα προγράμματα υποδομών αντίστοιχα με αυτά ε, της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί μιλήσαμε για διάφορα προγράμματα στη Βιέννη, στην Βρατισλάβα, Ρουμανία, Βουλγαρία για να αυξηθεί η διασύνδεση μεταξύ των περιφερειών. Θα υπάρχουν αντίστοιχα προγράμματα και στο μέλλον. Κύριε Επίτροπε, παρακαλώ να είστε σύντομος. Ευχαριστώ σε την αφορά Δεν μπορώ να σας δώσω μια συγκεκριμένη απάντηση γιατί αυτό διαφέρει ανάλογα με την κάθε περιφέρεια, αλλά και εντό τη κάθε περιφέρεια υπάρχουν ε, αποκλήσεις. Αλλά εκείνο που μπορούμε να παρατηρήσουμε συνολικά είναι ότι ε, τα έργα στον χώρο της ε, έρευνας και της καινοτομίας έχουν ψηλότερη ζήτηση και ειδικότερα έργα τα οποία αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό σας λέω τώρα συνολικά. Υπάρχουν διαφορές σε ό,τι αφορά τα επιμέρους ε, κράτη-μέλη. Ε, σε ό,τι αφορά την έκθεση Πάρκα, ε, έχω ζητήσει από τον Μαρίτσια που και σε ευχαριστώ Ντανούτα που ανακάλυψες αυτή την έκθεση. Εγώ θα συνεχίσω να τον απασχολώ ως σύμβουλό μας ούτως ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και σε σχέση με αυτή την έκθεση. Για να δούμε τι μπορούν να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα έχουμε στο μέλλον και διασκέψεις με stakeholders, με εμπλεκόμενους ε, φορείς ε, και θα υπάρξουν και συμφωνίε στο πλαίσιο αυτών των διασκέψεων. Μετά, σε ό,τι αφορά την ε, περιφέρεια, την περιοχή του Ντούναβη, υπάρχουν προτάσεις για κοινού στόχου και γι' αυτό έγινε και η πρόταση για την εκπόνηση μια κοινή στρατηγικής η οποία θα εστιάζει σε ορισμένα κύρια ζητήματα, ούτω ώστε να μην συμπεριληφθούν εδώ τα πάντα και να πλατιάσει υπερβολικά μια τέτοια πολιτική. Ε, και για να μην συμβεί αυτό που είπα, δηλαδή περιφερειακά προβλήματα περιφερειακής φύσης δεν μπορούν να επιληθούν με τη μετάθεση του στο μακροπεριφερειακό επίπεδο. Όμως ε, το ε, λέμε ξανά και ξανά πως θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ περιφερειακού και μακροπεριφερειακού επίπεδου ούτως ώστε να είναι δυνατή η ευκολότερη επίλυση διμερών προβλημάτων από ότι σε, αυτό θα συνέβαινε σε μια αμυγός ε, διμερή σχέση. Ε, κύριε Ομπέμα, σε ό,τι αφορά ε, τις χώρες εκείνες με προβλήματα, με λιματικούς προπολογισμούς, ε, δεν σας είπα ε, πώς θα πρέπει να λάβει η χώρα εδώ μια αυξημένη χρηματοδότηση, ένα αυξημένος προπολογισμός, απλά είπα ότι η διαρθρωτική χρηματοδότηση θα πρέπει να συνεχιστεί όπως αυτό συνέβαινε μέχρι τώρα δηλαδή υποβολή έργων, προγραμμάτων, απορρόφηση, δέσμευση, commitment, δηλαδή ό,τι κάναμε μέχρι τώρα. Και προφανώς στο πλαίσιο της ε, πολιτικής ε, συνοχής υπάρχουν ε, δυνατότητες για να παρέμει κανείς σε ό,τι αφορά τέτοιες ε, περιπτώσεις ε, χωρών δηλαδή με ελληματικούς αλλά εγώ εξακολουθώ να θεωρώ πως αυτά τα κονδύλια της περιφερειακής πολιτικής θα πρέπει να αξιοποιούνται για να δίνεται οικονομική όθηση στις ε, ε, στις ε, περιφέρειες αλλά δεν θέλω να δοθεί εντύπωση πως αυτοί που δημιουργούν αυτά τα προβλήματα που έχουν αυτά τα προβλήματα με τους προπολογισμού θα πρέπει να ε, λάβουν και έπαινο για αυτό που έκαναν απλά είπα ότι δεν θα πρέπει να μπερδεύουμε το ένα με το άλλο σε ό,τι αφορά την περιφερειακή συνοχή την εδαφική σύνομη, ε, ε, πολιτική και συνοχή. Προφανώς υπάρχει εδώ ε, μια αύξηση σε ό,τι αφορά την, το ρυθμό της απορρόφησης Τώρα, ε, σε, σε, κύριε, ε, αυτό που αναφέρεται κύριε ε, δηλαδή στην συγχρηματοδότηση, προφανώς ναι, είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται αυτή η συγχρηματοδότηση, αλλά από εκεί και μετά έχει αναλυθεί η δέσμευση από την πλευρά των κρατών μελών να γίνεται επιπρόσθετη, αν θέλετε, χρηματοδότηση, που δεν σχετίζεται μια τέτοια επιπρόσθετη χρηματοδότηση με τη συγχρηματοδότηση. Και να πούμε πως ε, εκ των ε, προτέρων ήμασταν πολύ ε, φιλόδοξοι γιατί τώρα με βάση την οικονομική κρίση δεν νομίζω πως θα λάβουν χώρα τέτοιες προσθέτες ε, χρηματοδοτήσεις. Ε, σε ό,τι αφορά την έκθεση της ε, Επιτροπής, ναι, έχουμε τα συγκεκριμένα simplification packages, αυτές δηλαδή τις προτάσεις για απλούστευση των σχετικών μέτρων και μέσα σε αυτή την περίοδο έχουμε ήδη λάβει τα σχετικά μέτρα και μένει να δούμε κατά πόσο θα λειτουργήσει κάτι τέτοιο αναφέρεται και από άλλους συναδέλφους ότι η κοινωνική πτυχή θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί ε, τμήμα της ε, πολιτικής μας ε, συνοχής και προφανώς η έκθεση για την πολιτική συνοχής θα πρέπει να δίνει κάποια στοιχεία σε ό,τι αφορά τη μελλοντική ε, χάραξη της πολιτικής. Αλλά καταρχήν πρόκειται, δηλαδή με αυτό, ε, σε ό,τι αφορά αυτό το κείμενο, για κάποιες αρχικές ε, προτάσεις, οι οποίες θα συζητηθούν περαιτέρω, με βάση ένα μια πραγματιστική προσέγγιση σε ό,τι αφορά το τελευταίο ερώτημα, σε ό,τι αφορά δηλαδή τα τρένα ε, μεγάλης αυτό δεν αποτελεί κάτι το οποίο μπορεί να κινήσει η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό εξαρτάται ακριβώς από το επίπεδο των μακροπεριφερειών και της ε, ε μεγαλύτερης απόδοσης, δηλαδή αυτό που είπα προηγουμένως, όντως ώστε να έχουμε ε, ένα έργο το οποίο θα λαμβάνει η χώρα ταυτόχρονα σε διαφορετικά κράτη-μέρη, σε διαφορετικέ περιφέρειε, ώστε να μην έχουμε για παράδειγμα ένα τρένο υψηλή ταχύτητα το οποίο θα αρχίσει κάπου, όλα. δεν θα φτάνει κάπου. Αγαπητοί συνάδελφοι, άλλοι οκτώ έχουν ζητήσει το λόγο. Θα ήθελα αυτοί που μπορούν να πούν ότι δεν θα μιλήσουν να το κάνουν. Αν κάποιοι επιμένετε όχι πάνω από μισό λεπτό. Τα τρία ερωτήματά μου αφορούν την ε, αστική ανάπτυξη και την περιφερειακή ανάπτυξη. Ε, το 1999-2006 με το 6 ε, είχαμε ένα ε, πρώτο πρόγραμμα το οποίο δεν ήταν τόσο χρήσιμο αλλά είχαμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα και αυτά τα συμπεράσματα θέλαμε να έχουν ενσωματωθεί μέσα στη νέα προγραμματική περίοδο σε ό,τι αφορά δηλαδή την οικονομία, την οικολογία και ούτω καθεξής. Ε, αυτό όμως δεν συνέβη στις περισσότερες περιφέρειες να ληφθούν δηλαδή υπόψη αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή ε, τι νόημα έχει να έχουμε ένα τέτοιο ακριβό ε, πείραμα το οποίο μας οδηγεί σε κάποια συμπεράσματα το οποίο όμως δεν λαμβάνουμε υπόψη μας. Άρα λοιπόν αυτό το mainstream, αυτή η ένταξη στις πολιτικές που εφαρμόζονται σε ό,τι αφορά αυτά τα έργα θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Δεύτερο ερώτηση, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία εντός των ίδιων των κρατών μελών. Έχουμε την διαπαθή, αν θέλετε των ε, πρωτευουσών με τις ε, πιο απομακρυσμένες περιοχές. Εσείς ε, πώς μπορείτε μια κοινωνική πρωτοβουλία να έχετε κάτι το οποίο θα εστιάζει περισσότερο στην διαπεριφερειακή συνεργασία παρά τη συνεργασία περιφερειών με την πρωτεύουσα. Από εκεί και μετά πώς μπορούμε να κινηθούμε πέρα από τις περιφέρειες όπως αυτές από αυτές τις περιφέρειες όπως τις ορίζουμε ε, μέχρι τώρα. Δηλαδή, εγώ προέρχομαι από μια περιφέρεια της Γερμανίας όπου έχουμε 2,3 εκατομμύρια πολίτες και εντασσόμαστε σε μια κοινή ε, περιφέρεια, με δύο άλλα ομόσπονδα κρατήδια. Με αποτέλεσμα η συνεργασία μεταξύ μας είναι δυσκολότερη από ότι η συνεργασία με περιφέρεια άλλου κράτους Τι θα κάνουμε στην ουσία με αυτό. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε και σας ευχαριστούμε θερμά που αμέσως μετά την καταιγίδα σπεύσατε να επισκεφτείτε τη Γαλλία. Το εκτίμησε ιδιαίτερα ο τοπικός πληθυσμός αλλά και ολόκληρη η Γαλλία. Δεν κατάλαβα την απάντησή σας για τα προγράμματα έρασμος των τοπικών και περιφερειακών αντιπροσώπων. Το 2008 είχαμε μια καταπληκτική έκθεση ό,τι αφορά τα πλεονεκτήματα του έρασμο για τους τοπικούς και περιφερειακούς αντιπροσώπους και μάλιστα είχε γίνει ενθουσιοδός δεκτή αυτή η έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας είχα στείλει και επιστολή τότε και μου απαντήσατε ότι μια, συμβουλευτική, μια εταιρεία συμβουλών, Εκοτέ και Κορίς, ασχολούνται με την ανάλυση και την αξιολόγηση της πολιτικής αυτής ε, για τη σκοπιμότητα συνέχισής της και ότι τα πρώτα στοιχεία της ανάλυσης αυτής ήταν μάλλον θετικά για την ε, συνέχιση του έρασμος. Τι συμβαίνει σήμερα. Ποια είναι η προοπτική κατά τη γνώμη σας για το έρασμος, για τους τοπικούς και περιφερειακούς αντιπροσώπους, γιατί είναι πολύ σημαντικό και έχει τεράστια πλεονεκτήματα αυτό το πρόγραμμα. Σε ό,τι αφορά την πολιτική για τις πόλεις, είπατε στην ακρόασή σας ότι στόχος σας είναι να εφαρμοστεί μια αυθεντική πολιτική για τις πόλεις. Έχει περάσει κάποιος χρόνος από τότε που αναλάβατε τα καθήκοντά σας. Ποιοι θα είναι κατά τη γνώμη σας οι βασικοί άξονες αυτής της πολιτικής για τις πόλεις. Και μία ευαισθητοποίηση. Για 15 χρόνια εφαρμόστηκε στην Γαλλία η πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης με τα διαρθρωτικά ταμεία. Σας διαβεβαιώ ότι η πολιτική αυτή έχει απτά αποτελέσματα και συγκεκριμενοποιεί την κοινοτική παρέμβαση στις διάφορες περιφέρειες και φέρνει τους πολίτες πολύ πιο κοντά στην Ένωση εξαιτίας ακριβώς αυτών των απτών αποτελεσμάτων. Είναι βέβαια περίπλοκη η εφαρμογή αυτής της πολιτικής, γι' αυτό και η εικόνα που δίνει είναι μερικές φορές δυσνόητη. Γιατί είναι περίπλοκο όλα αυτά τα ντοσιά για τα διαρθρωτικά ταμεία. Και μερικές φορές είναι αντιπαραγωγική εικόνα που δίνει η περιφερειακή πολιτική, παρόλο που η ουσία της είναι πολύ θετική. Είπατε ότι χρειάζεται διαφάνεια αλλά δεν θα πρέπει να είμαστε υπερβολικοί στους ελέγχους, γιατί η πληθώρα ελέγχων σκοτώνει τη δράση και οι υπερβολικές διατυπώσεις και γραφειοκρατία διακυβεύουν την θετική εικόνα που είχε μέχρι στιγμής η περιφερειακή πολιτική στις ε, ευρωπαϊκές περιφέρειες. Η κυρία Κάντεμπαχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Θα συμφωνήσω με τα όσα είπε. Ε, αυτό που χρειαζόμαστε στην ε, πολιτική ε, συνοχή είναι ένα καλύτερο marketing. Νομίζω πως όλοι μας εδώ γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η πολιτική συνοχή, αλλά όταν ρωτάμε τις θέσεις περιφέρειες τι ακριβώς συνιστά αυτή η πολιτική δεν έχουν να μας δώσουν μια συγκεκριμένη απάντηση. Και βέβαια αντιλαμβάνομαι ότι γίνεται συχνά, συναδελφοί προσπαθούν έτσι να παρουσιάσουν αυτές τις επιτυχίες ως δικές τους με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μια συγκεκριμένη αντίληψη ε, των πολιτών ε, ε, της Ευρώπης σε ό,τι αφορά αυτή την πολιτική συνοχή. Και ε, θα πρέπει να αυξηθεί ακριβώς αυτή η ορατότητα αυτής της πολιτικής ούτως ώστε να παραμένει και η βούληση από την πλευρά των πολιτών των κρατών μελών εκείνων τα οποία κυρίως ε, ε, συνεισφέρουν περισσότερο χρηματοδοτικά ούτως ώστε λοιπόν η άποψή τους να είναι πιο θετική ούτως ώστε να αντιλαμβανόμαστε ότι δεν πρόκειται απλά για ένα sponsoring εδώ αλλά πρόκειται για μια επένδυση από την οποία τελικά αποκομίζουν κάτι όλοι οι πολίτες της Ευρώπης. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτό το πέρα από τα, τα τρία, τις τρεις τεχνικές αρχές, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της πολιτικής, θα πρέπει να έχουμε και την αρχή αυτή του marketing, ούτως ώστε να καταστεί σαφής ε, η πολιτική και η λογική που ακολουθεί με αυτή την ε, πολιτική. Ε, you are not here, I understand. Uh, Josip Matula, please. Yes, I'm sorry. Yeah. I'm sorry. Yeah. Ε, ε, ναι, Οι διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκονται στο τελικό στάδιο της Εμπορική συμφωνίας με την Κολομβία και το Περού. Η συμφωνία αυτή θα θίξει τις υπερπεριφέρειες σε εισαγωγικά της Καραϊβικής. Η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θυσιάζει τους κατοίκους και τους οικονομικούς εμπλεκομένους στην περιοχή αυτή. Δύο ερωτήσεις λοιπόν. Τι νόημα έχει να υπάρχει μια στρατηγική για το 2020 αν δεν υπάρχει μια συνοχή στα μέτρα τα οποία θα λαμβάνονται. Δεύτερη ερώτηση. Η ανακοίνωσή σας περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία σε ποιο βαθμό θα ληφθούν υπόψη. Σας ευχαριστώ. Μία ερώτηση έχω μόνο που θα είναι πολύ συνοπτική. Εμείς οι Ευρωβουλευτές πολύ συχνά μεταφέρουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών αλλά και τις επικρίσεις που ακούμε πολλές φορές. Έχουμε αγαστή συνεργασία μέχρι στιγμής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό θα ήθελα να σας υποβάλω μία ερώτηση. Οι δικές σας προσδοκίες ποιες είναι τι περιμένετε εσείς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ευελιξία, την ελαστικότητα, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των διαρθρωτικών ταμείων. Ο κύριος Ρικάρδο Κορτές Λάστρα. Η πολιτική συνοχή, κύριε Επίτροπε, είναι ακρογωνία ως λήθος της ευρωπαϊκής πολιτικής. Μια πολιτική που έχει μέσο και μακροπρόθεσμη διάσταση. Το δικό μου μήνυμα είναι ότι είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής είναι να θέσει στο επίκεντρο της στρατηγικής του 2020 την πολιτική συνοχής. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μέσω της πολιτικής συνοχής οικοδομούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και θα πρέπει να εμπλέξουμε και τις ε, περιφερειακές και τοπικές αρχές στη διαμόρφωση αυτής της πολιτικής συνοχής. Έχω και μία ερώτηση. Ποιοι, κατά τη γνώμη σας, είναι οι μηχανισμοί για να ενισχύσουμε την ε, συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών ε, αρχών στην οικοδόμηση της Ευρώπης. Κύριε Επίτροπε, λέει ο κύριος Τεϊσέρα, είπατε στις εισαγωγικές σας ομιλίες ότι ο στόχος της περιφερειακής πολιτικής δεν είναι μόνο να απομίζει κονδύλια, αλλά να χρηματοδοτεί και να εφαρμόζει βιώσιμα προγράμματα και σχέδια. Σας συγχαίρω και για την ε, άμεση αντίδρασή σας ως προς την καταστροφή και τη θεμηνίες στη Μαδέρα του Φεβρουαρίου. Βέβαια, δεν φταίει μόνο η νομοθεσία, αλλά σίγουρα για να δρομολογηθούν γρήγορα οι ενισχύσεις προς τη Μαδέρα θα πρέπει να περιοριστεί η γραφειοκρατία. Την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή η Πορτογαλία υπέβαλε οριστικά ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη, την αποτίμηση της καταστροφής που είναι 1 δισεκατομμύριο 80 εκατομμύρια. Στην περίοδο προγραμματισμού 2000-2006 είχαμε λάβει 1 δισεκατομμύριο 98 εκατομμύρια και μέσα σε 6 ώρες ε, καταστράφηκαν ουσιαστικά σχεδόν όλα, όλες οι κοινωτικές επενδύσεις στη Μαδέρα γιατί ήταν περίπου η αποτίμηση των ζημιών ε, τόσο όσο είχαμε λάβει στην ε, περίοδο 2000-2006. Ε, Από το 1 δισεκατομμύριο, 80 εκατομμύρια που ήταν οι ζημιές στη Μαδέρα θα χρειαστούν τεράστιες ενισχύσεις για την ανοικοδόμηση. 740 εκατομμύρια θα δώσει η πορτογαλική κυβέρνηση ο τοπικός προϋπολογισμός της Μαδέρας ε, θα προσφέρει περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ, οπότε αυτό που περιμένουμε από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ταμείο Αλληλεγγύης είναι μόνο 30 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει τεράστια δυσαναλογία μεταξύ του ύψους των ζημιών και της ε, προσφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης προς τη Μαδέρα. Δεν πιστεύετε ότι είναι τεράστια αυτή η δυσαναλογία και πολύ άδικη. Δεν είναι κατάλληλη ώρα, κύριε Επίτροπε, ώστε μαζί με τους ε, συναδέλφους σας να σκεφτείτε σοβαρά την ανάγκη αναθεώρησης του Ταμείου Αλληλεγγύης. Γιατί είναι άλλη πραγματικότητα στις υπεραπόμακρες περιοχές. Εκεί είναι τεράστιοι περιορισμοί και οι κλιματικές αλλαγές και οι κλιματικές ε, συνθήκες πολλές φορές ε, δυσχεραίνουν την κατάσταση. Δεν πρέπει το Ταμείο Αλληλεγγύης να γίνει πιο ελαστικό, η κινητοποίησή του να γίνεται πιο άμεση, και να αποφεύγονται οι καθυστερήσει, γιατί έχει μπλοκάρει αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιστεύω ότι είναι προ όφελο όλων και αυτών που δεινοπάθησαν, αλλά και αυτών που στο μέλλον θα υποστούν ε, τι θεομηνίε. Καλό θα ήταν από τώρα, κύριο Επίτροπο, μαζί με του συναδέλφου του να εγγύψει αυτό το θέμα τη αναθεώρηση του Ταμείου Αλληλεγγύη. Κύριε Επίτροπο, έχετε το λόγο για τι τελευταίε απαντήσει. Ε, Ευχαριστώ σε ό,τι αφορά όλο το ζήτημα αυτών των πόλεων, μετροπόλεων ε, και τη σχέση με τις περιφέρειες. Ε, πράγματι είναι ένα αρκετά περίπλοκο ζήτημα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Είναι πολύ ε, σύνθετα εδώ τα ζητήματα. Υπάρχουν μικρές, μεγαλύτερες πόλεις, πρωτεύουσες και ούτω καθεξής. Πρόκειται λοιπόν για έναν περίπλοκο τομέα ε, πράγματι είχατε δίκιο σε αυτό που αναφερθήκατε, δηλαδή με τα διάφορα προγράμματα ε, κάναμε εδώ κάποιες πολύ συγκεκριμένες ε, παρατηρήσεις και είδαμε ότι στο πλαίσιο του management, θέλετε, από την πλευρά των περιφερειών, πολλά από αυτά τα συμπεράσματα δεν αξιοποιήθηκαν. Ενώ υπήρξαν κάποιοι όπως το Ολλανδία και το Ρότερνταμ που έλαβαν υπόψη τους αυτά τα συμπεράσματα, δηλαδή όπου υπήρχε μια κοινή συμπερίληψη. Ε, ε, θα πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν το ε, πώς μπορούμε να έχουμε ακριβώς αυτή την προσαρμογή χωρίς να δημιουργηθούν επιπρόσθετα προγράμματα. Το θετικό γεγονό ήταν ακριβώς αυτό ότι μπορούσαμε να μειώσουμε τον αριθμό των διαφορετικών έργων, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να δίνεται η έμφαση στα σημεία που χρειάζεται. Αυτή είναι και η πρόκληση από εκεί και μετά σε ό,τι αφορά την διαπεριφερειακή συνεργασία εντό τη επικράτειας ενό ε, και μόνο κράτου μέλου, ε, θα πρέπει να σα πω ότι θα πρέπει να το το καλύτερο αυτό το ζήτημα. Ε, πολλά ζητήματα δεν μπορούν να επιληθούν με την προσέγγιση top-down, δηλαδή από τα πάνω προ τα κάτω. Εκεί χρειάζεται συνεργασία μεταξύ των ίδιων των περιφερειών με την βοήθεια των, του ανώτερου, αν θέλετε, επίπεδου. σίγουρα χρειάζονται κάποιες ε, επιπρόσθετες ε, απλουστεύσεις σε ό,τι αφορά το ένα ή το άλλο επίπεδο συνεργασίας. Τώρα, ε, σε ό,τι αφορά, τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή και τον θα έχουμε την, μια σχετική συζήτηση, αλλά δική μου άποψη είναι πως θεωρώ πάρα πολύ λογικό, πάρα πολύ χρήσιμο ε, και σκόπιμο ένα τέτοιο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργήσει και οι σχετικές εμπειρίες που έχουμε σε αυτό το τομέα θα πρέπει πράγματι να αξιοποιήσουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα το τομέα του marketing και της παρουσίασης, η αρμόδια ε, μονάδα της Γενικής Διεύθυνσης ε, έχει εκπονήσει μια, ένα σχετικό έγγραφο το οποίο καλύπτει τα πλέον σημαντικά έργα σε ό,τι αφορά τις ε, περιφέρειες των ευημέρους ε, κρατών ε, μελών. Πρόκειται για ένα αντίγραφο το οποίο μπορείτε να λάβετε και εσείς ούτε ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για την παρουσίαση της πολιτικής γιατί πράγματι μπορεί να αποτελέσει κάτι το χρήσιμο σε ό,τι αφορά το marketing από τη μέσα πλευρά και εδώ να περάσω ε, στο ζήτημα των προσδοκιών απέναντι στους ε, ευρωβουλευτές. Εδώ το ζητούμενο είναι εδώ στις Βρυξέλλες και ε, στο Στρασβούργο με βάση δηλαδή τη δικτύωση που έχετε να διασφαλίσετε ότι θα τηρήσει το ίδιο επίπεδο το οποίο έχει διασφαλίσει μέχρι τώρα η περιφερειακή πολιτική και από εκεί και μετά να εξελιχθεί με κάποιους ε, τρόπους και ταυτόχρονα να ε, διασφαλίζεται και η κατάλληλη εφαρμογή των σχετικών έργων της ε, πολιτικής αυτής στα επιμέρους κράτη-μέλη. Αυτό το υπενθυμίσουμε και πάντοτε στις εθνικές ε, κυβερνήσεις και στους εθνικούς αρμόδιους όπου υπάρχουν ελλείψεις θα πρέπει να γίνονται ε, απαραίτητες διορθώσεις σε ό,τι αφορά το επόμενο ζητήμα που θέσατε θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε διμερώς αλλά αν δείτε και την ε, επόμενη περίοδο την χρηματοδοτική πράγματι υπάρχουν και κάποιες και κάποιες ε, προβλέψεις και στην ε, Λισαβόνα κάποιες ε, σαφείς αναφορές σε ό,τι αφορά τις ε, ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές όπου τονίζεται ακριβώς η ιδιαίτερη σημασία και ο ευαίσθητος χαρακτήρας των πλέον απομακρυσμένων περιφερειών. σε ό,τι αφορά τώρα τα βοηθητικά έργα Πρόκειται για ένα περίπλοκο ζήτημα, χρειάζεται εδώ να γίνει μια ιδιαίτερη συζήτηση. Υπάρχει μια πρόταση που είχε γίνει για σχετική νομοθετική τροποποίηση το 2005 που είχε συγκεντρώσει μάλιστα και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά όχι του Συμβουλίου. Εγώ ξαναήρθα σε επαφή με την Ισπανική Προεδρία για το ενδεχόμενο μια νέα προσπάθεια, μια νέα πρωτοβουλία με κάποιε τροποποίησει. Αλλά σε ό,τι αφορά τον πυρήνα, αν θέλετε, η αλληλεγγύη εδώ δεν ε, σημαίνει ότι ε, μπορούμε να έχουμε πάντα υποκατάσταση από το ένα εργαλείο στο άλλο, αλλά συζητάω ήδη με την ε, που του ότι θα μπορούσαμε ενδεχομένω να έχουμε ένα κοινά εργαλεία τα οποία θα υπάρχουν διαθέσιμα αλλά το Ταμείο συνεχίζει από εκεί και μετά προβλέπεται για την ε, ανάκαμψη και βέβαια αυτό εξηγεί εν μέρη και το γιατί πολλέ φορέ υπάρχουν καθυστερήσει, γιατί χρειαζόμαστε δηλαδή τη σύμφωνη γνώμη από την πλευρά του Κοινοβουλίου και από την πλευρά του Συμβουλίου ε, σε ό,τι αφορά την ε, κατανομή των σχετικών κοντιλίων. Δεν μπορώ να απαντήσω άμεσα σε αυτό το ερώτημα που θέσατε, αλλά είχα την την ευκαιρία να συναντηθώ με τον πρόεδρο Σατίν, ο οποίος μου είπε πως η κατανομή αλλά και η απορρόφηση στην Πορτογαλία λαμβάνει ε, χώρα με πολύ καλό τρόπο και βλέπουμε πράγματι να εφαρμόζεται και μια ε, ευελιξία εδώ και από εκεί και μετά το κατά πόσο ε, μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτό το είδος governance στο οποίο αναφερθήκατε παραμένει πάντα ένα ζήτημα ανοιχτό γιατί ε, από την πλευρά των περιφερειών θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι συμμετέχουν, ότι εμπλέκονται μέσα στον ε, σχεδιασμό των επιχειρησιακών προγραμμάτων πράγμα το οποίο βέβαια δεν αφορά μόνο τις περιφέρειες αλλά και τα επίπεδα που βρίσκονται κάτω από τις περιφέρειες αυτές. Ε, και εδώ έχουμε να θυμίζουμε και την έκθεση αλλά και τη λευκή ε, βίβλο που έχει εκπονήσει σχετικά η Επιτροπή των Περιφερειών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι εκπροσωπώ όλους συναδέλφους εδώ ε, λέγοντα ότι ήταν πολύ καρποφόρα η ανταλλαγή απόψεων, οι απαντήσεις πολύ εμπεριστατωμένες και πολύ διεξοδικές ε, και φαντάζομαι είδατε ότι μας είστε ιδιαίτερα συμπαθείς και μπορείτε να υπολογίζετε στην υποστήριξη της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν πρόκειται να γίνει διάλειμμα τώρα. Όσοι πρέπει να φύγουν, να το κάνουν παρακαλώ χωρίς μεγάλη φασαρία. Θα πρέπει να περάσουμε στο σημείο 5. Ελπίζω να έχει παραμείνει στην αίθουσα η Ραμόνα Μανέσκου, γιατί προβλέπεται μια μήνυα ακρόαση στα πλαίσια του εγγράφου εργασία ε, της κυρίας Ραμόνα Μανέσκου. Αν θέλετε κάντε μας μια σύντομη εισαγωγή και μετά θα περάσουμε στην ακρόαση. Ελπίζω να έχουν έρθει όλοι οι προσκεκλημένοι μας για να αρχίσει η ακρόαση που οργάνωσε η κυρία Μανέσκου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχουμε καθυστερήσει κάπως, γι' αυτό και θα παρουσιάσω τηλεγραφικά τα έγγραφα εργασία μου που αφορά τη χρηστή διακυβέρνηση θα σας πω λίγα λόγια για το έγγραφο εργασίας μου που απαρτίζεται από δύο τμήματα. Ένα τμήμα που αναλύει τη Λευκή Βίβλο για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και εγκρίθηκε πέρυσι τον Ιούλιο και το δεύτερο τμήμα που επιχειρεί μία εξέταση των μηχανισμών διαχείρισης και των ε, ευθυνών που επιρρύπτονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αφενό και στα κράτη-μέλη αφετέρου. Σε ό,τι αφορά το πρώτο τμήμα της έκθεση μου, του εγγράφου εργασία, όπως σας είπα, προβαίνει σε μια σειρά αξιολογήσεων και συστάσεων στα πλαίσια της ανάλυση που προβαίνει για τη Λευκή Βίβλο. Έχω μερικές πολύ σημαντικές συστάσεις ως προς το θέμα της ε, χρηστής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα των δύο διαστάσεων της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, της κάθετης κατακόρυφης και της οριζόντιας διάστασης. Σίγουρα υπάρχουν πολλά επίπεδα διακυβέρνησης. Είναι σημαντικό λοιπόν να εξασφαλίσουμε την συνεργασία και σε κάθετο επίπεδο μεταξύ του κράτους και των τοπικών αρχών, αλλά και σε οριζόντιο επίπεδο μεταξύ των διαφόρων φορέων της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο προβλέπει την ανάγκη ορισμού της αρχής της εταιρικής σχέσης. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θεσμοθετημένος ορισμός της εταιρική σχέση. Θα πρέπει λοιπόν να καταρτήσουμε, να θεσπίσουμε έναν ορισμό και να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε εταιρική σχέση. Κάτι που προϋποθέτει φυσικά την εφαρμογή γνήσεων εταιρικών σχέσεων μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Πολύ σημαντική είναι η εξασφάλιση μόνιμου διαλόγου μεταξύ των τοπικών αρχών ήδη από την έναρξη των διαπραγματεύσεων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει επίσης να εκμεταλλευτούμε και να αξιοποιήσουμε καλύτερα την εδαφική συνοχή και η συμμετοχή των υποεθνικών παραγόντων στην υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή της εδαφικής συνοχής. αλλά και η εδαφική συνεργασία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της στρατηγικής του 2020. Κάτι που έχει υπογραμμιστεί σε πολλές απαντήσεις που δόθηκαν κατά την πρόσφατη δημόσια διαβούλευση. Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας, αλλά και οι διάφορες εταιρικέ σχέσεις ε, και εμπειρίες που στηρίχθηκαν στα προγράμματα Urban και Leader, θα πρέπει να προωθηθούν ως μέσα οργάνωσης συστημάτων διασυνοριακής διακυβέρνησης και διασφάλισης της ιδιοκτησίας των διαφόρων πολιτικών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ένα άλλο σημαντικό θέμα αφορά την απλούστευση των κανόνων σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, που αποτελεί προϋπόθεση για την καλύτερη διακυβέρνηση κατά την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Οι πρόσφατες μάλιστα τροποποίησεις των γενικών διατάξεων ε, και του κανονισμού του ΦΕΝΤΕΡ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, είναι σημαντικά βήματα πρόοδου Βέβαια, δεν θα πρέπει η απλούστευση των κανόνων να έχει προσωρινό χαρακτήρα εξαιτία της οικονομικής χρήσης. Θα πρέπει να μονιμοποιηθούν αυτοί οι κανόνες απλούστευσης. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε και το πρόγραμμα Έρασμος για τους τοπικούς και περιφερειακούς αντιπροσώπους, όπως υπογράμμισε και στην ομιλία μου προς τον Επίτροπο, θα πρέπει να υποστηρίξουμε τη συνέχιση αυτού του προγράμματος και να προβλέψουμε επαρκή χρηματοδότηση στο πλαίσιο των προσεχών διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να ενισχύσουμε τη δικτύωση με τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές. Καλό θα ήταν να ανακαταρτήσουμε και ένα χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση γιατί ένα τέτοιο μέσο θα είναι πολύ πρόσφορο για την ανάπτυξη μιας κοινή προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης. Το δεύτερο τμήμα του εγγράφου εργασίας μου εξετάζει τους μηχανισμούς ελέγχου και αναζητά κάποιες λύσεις για τη βελτίωση των υφισταμένων μηχανισμών ελέγχου εφαρμογής των προγραμμάτων. Ε, η παρακολούθηση που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή είναι ανεπαρκής. και δεν αρκεί για να συμπληρώσει τους ανεπαρκείς ελέγχους που γίνονται και στα κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι και στη, κατά τη φάση, την αναρκτήρια φάση των προγραμμάτων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να έχει ενισχυμένο ελεγκτικό ρόλο. Και ο ενισχυμένος αυτός ε, ελεκτικός ρόλος θα πρέπει να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος. Επίσης ε, θα πρέπει να προβλέπονται ad hoc ε, έλεγχοι και συντονισμός με τις τοπικές ελεκτικέ αρχές προκειμένου να διορθωθούν οι παρατυπίες και οι ατασταλίες και να περιοριστεί το περιθώριο λάθος. Επίσης, η έρευνα θα πρέπει να εντοπιστεί στο επίπεδο που διαπράττονται τα περισσότερα σφάλματα και κυρίως στις μη επιλέξιμες δαπάνες αλλά και στις δημόσιες προμήθειες. Γιατί σε αυτούς τους δύο τομείς εντοπίζουμε τις περισσότερες παρατυπίες και ατασταλίες. Επαναλαμβάνω ότι υπέρ της απλούστευσης των κανόνων ώστε να γίνουν πιο προσιτές ε, οι διαδικασίες για τους ενδιαφερόμενους και να μην αποθαρρύνονται οι επίδοξοι δικαιούχοι των σχεδίων από την υπερβολική γραφειοκρατία. Εκτός από τα προγράμματα και τα σχέδια θα πρέπει να ενισχύσουμε και τη συνδρομή που παρέχει η Επιτροπή στις διαχειριστικές αρχές δεδομένου ότι τα περισσότερα σφάλματα εμφανίζονται σε επίπεδο πρωτοβάθμιου ελέγχου. Επίσης, απαιτείται ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων επιπέδων ελέγχου για να αποφευχθεί ο υπερβολικός έλεγχος ή ο διπλός έλεγχος. οι μηχανισμοί Jeremy και Jaspers θα πρέπει να αξιοποιηθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω οι δυνατότητέ του, προκειμένου να καταστεί δυνατή και η ανάπτυξη ποιοτικών στρατηγικών προγραμμάτων και η συμμετοχή ιδιωτικών φορέων και κεφαλαίων στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Βέβαια, οι τοπικοί και περιφερειακοί εκπρόσωποι μίλησαν για την ανάγκη μεγαλύτερου συντονισμού, μεγαλύτερης ελαστικότητας των ταμείων και μιας ανάγκης ολοκληρωμένης προσέγγισης, καθώς και βελτίωσης της συνεκτικότητας των κανόνων. Αυτά προς το παρόν και περιμένω τους προσκεκλημένους εμπειρογνώμενους. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Έχουμε τρεις φιλοξενούμενους. Έχουν προσκληθεί από την κυρία Μανέσκου και οι τρεις. την κυρία Γκουρντά, την κυρία Γκούναρσον και τον κύριο Λουκ Χέντριξ από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα ήθελα να σας ζητήσω να είστε σύντομοι να μην ξεπεράσει ο καθένα τα 10 λεπτά. Θα πρέπει να ξεκινήσω με την κυρία Γκουρντά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εξαιτίας της κυρίας Μαριάνου, η, τη Γενική Διευθύντρια δηλαδή, η οποία δεν μπόρεσε να είναι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ επίσης την κυρία Μανέσκου γιατί δίνει την δυνατότητα στην οργάνωσή μας να πάρει το λόγο εδώ. Θα ήθελα να σας μεταφέρω αυτά τα οποία είχε προετοιμάσει η κυρία Μαριανού. Η διάσκεψη των περιφερειών της Ευρώπης συγκεντρώνει 160 περιφερειακές αρχές από κράτη-μέλη της Ένωσης αλλά και των χωρών γειτονίας. Είναι μια οργάνωση 37 ετών σήμερα και η οποία όλα αυτά τα χρόνια προσπαθεί να προωθήσει τις περιφερειακές αρχές, να επηρεάσει τις κοινοτικές πολιτικές και να συγκεντρώσει την προσοχή στις επιπτώσεις που έχουν στις περιφερειακές πολιτικές τα κοινοτικά μέτρα. Τα τελευταία 20 χρόνια η δράση μας επέτρεψε να αλλάξει η εικόνα των περιφερειακών αρχών στην ευρωπαϊκή σκηνή. Σε μία πρώτη φάση είχαμε μία εικόνα θα έλεγα κάπως δευτερεύουσα. Στην ουσία δηλαδή ήμασταν εκεί μόνο και μόνο για να οικετεύουμε χρήματα από τα κοινοτικά όργανα, ενώ σήμερα ουσιαστικά οι πρωταγωνιστές είμαστε εμείς. Έχουμε την τεχνογνωσία, Ιδιαίτερα στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση και τον έλεγχο, ο πολλαπλασιασμός των εταίρων συνέβαλε στην ε, αύξηση του ελέγχου και στην περιπλοκή του έργου της αξιολόγησης. Βέβαια αυτός δεν είναι λόγος για να παλιδρομήσουμε και να υπαναχωρήσουμε σε σχέση με τους μηχανισμούς ε, διακυβέρνησης και μάλιστα δημοσιονομικής ε, και χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση ε, που χρειαστήκαμε χρόνια ολόκληρα για να του εφαρμόσουμε. Α μην ξεχνούμε ότι η ισχύ τη πολιτική αυτή ε, έγκυται στο ότι έχει φυγόκεντρη διάσταση. Πάει από το κέντρο προς τις περιφέρειες και έτσι γίνεται ορατή και στους πολίτες, ιδιαίτερα στην εποχή αυτή της κρίσης και της ε, αμφισβήτησης του ευρωπαϊκού οράματος. Γι' αυτό και η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλευρά των πολιτών είναι σήμερα σημαντικότερη από ποτέ. Πιστεύουμε επίση ότι η οικοδόμηση τη Ευρώπη, που είναι ένα sui generis οργανισμός, ένας ιδιότυπος οργανισμός, αντλεί τι δυνάμει τη από την εμπλοκή των περιφερειών και το γεγονό ότι γίνεται ο θεματοφύλακα των περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων και τη περιφερειακή πολυμορφία. Δεν θα πρέπει να ε, μετατρέψουμε την Ένωση σε ένα απλό οικονομικό χώρο απογυμνωμένο, πολιτικού περιεχομένου και απομακρυσμένο από τους πολίτες. Γιατί οι πολίτες είναι η ψυχή της Ευρώπης. Κατά τη γνώμη μας υπάρχει ένας κίνδυνος ε, συγκέντρωσης και πάλι της διαχείρισης της περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής των διαρθρωτικών ταμείων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί ίσως ε, μια συγκεντρωτική διαχείριση είναι είναι πιο απλή διαδικαστικά, αλλά έτσι απογυμνώνει την παρουσία της Ευρώπης από τις περιφέρειες. Και αυτό θα απομακρύνει ακόμη περισσότερο, θα αποξενώσει τους Ευρωπαίους πολίτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το νόημα που δίνουν σε αυτή την πολιτική. Θα πρέπει να δούμε τι μηχανισμοί υπάρχουν για τη διαχείριση της περιφερειακής πολιτικής σήμερα. Και φυσικά με απότερο στόχο την ε, όλο και πιο ενισχυμένη και ολοκληρωμένη Ευρώπη. Και υπό αυτό το πνεύμα υποβάλαμε κάποιε συστάσει ό,τι αφορά τη Λευκή Βίβλο για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη του 2009. Οι προτάσει μα στηρίζονται στην πολιτική αρχή που φέρει τον τίτλο Ευρωπαϊκό Εδαφικό Σύμφωνο που θα πρέπει να συναυθεί μεταξύ των Ευρωπαϊκών Εδαφών, των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το Ευρωπαϊκό, το Πανευρωπαϊκό Εδαφικό Σύμφωνο θα λάβει σάρκα και οστά μέσω δύο μηχανισμών. Ο πρώτος μηχανισμό είναι η σύναψη μια πολιτική συμφωνία για το όραμα, τους στόχους και τις προτεραιότητες της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Πρόκειται για μια συμφωνία που θα πρέπει να συναυθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλων των Ευρωπαϊκών Περιφερειακών Αρχών. Και μέσω αυτού του συμφώνου οι ευρωπαϊκές περιφέρειες αναλαμβάνουν τη δέσμευση να υλοποιήσουν την ευρωπαϊκή αυτή στρατηγική στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. Έτσι θα ενισχύσουμε την ιδιοκτησία της στρατηγικής αυτής από πλευράς ε, περιφερειών και θα γεφυρώσουμε το χάσμα που δημιουργήθηκε με τη στρατηγική της Λισαβόνας και θα υπερκεράσουμε τα εμπόδια, θα εξασφαλίσουμε εδώ και ένα καλύτερο συντονισμό στα διάφορα επίπεδα διαχείρισης, στο τοπικό, το περιφερειακό, το εθνικό και το υπερεθνικό, το κοινοτικό. Δεύτερος μηχανισμός ε, είναι η πολιτική συνοχής και η περιφερειακή πολιτική. Και εκεί πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δοθεί ένα συμβατικός χαρακτήρας στην εφαρμογή των πολιτικών αυτών με άμεση εμπλοκή και ανάμειξη των περιφερειακών αρχών, ανάλογα φυσικά με τις εθνικές ρυθμίσεις και θα μπορεί να έχει τη χαρακτήρα, δηλαδή τα συμβαλόμενα μέρη θα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι, οι τοπικές περιφέρειες ή θα έχει τριμερή χαρακτήρα με συμβαλόμενα μέρη την, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις περιφέρειες αλλά και τις εθνικές αρχές. Έτσι έχουμε δύο μηχανισμούς πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με τις στάσεις αυτές με πολλά πλεονεκτήματα. Τρία συγκεκριμένα. Το πρώτο πλεονέκτημα είναι ότι οι περιφέρειες αναλαμβάνουν ευθύνες, γιατί από τη στιγμή που αποκτήσουν ενοχικές συμβατικές ευθύνες, αποκτούν και νομικές ευθύνες και πολιτικές ευθύνες, οπότε θα αισθανιστεί καλύτερα μια περιοχή αυτούς τους στόχους και θα βάλει τα δυνατά της για να υλοποιήσει αυτούς τους στόχους, ευθυγραμμιζόμενοι με τους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα αυτή η υπευθυνοποίηση αποτελεί ένα βασικό μηχανισμό αμοιβέ εμπιστοσύνη που μπορεί να ισχύσει μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, των κρατών μελών και των υποεθνικών επιπέδων διακυβέρνηση. Το δεύτερο πλεονέκτημα είναι και το αρνητικό τμήμα, θα έλεγα, αυτό είναι το μοναδικό πράγμα, ο μοναδικός παράγον που θα μπορούσε να προκαλέσει την απλούστευση, την απλοποίηση. Η υπευθυνοποίηση των περιφερειακών και εθνικών εταίρων σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα κατά προτεραιότητα να δράσει σε στρατηγικούς άξονες μόνο και όχι να χαθεί στις λεπτομέρειες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα χάνει το χρόνο της σε διαδικασίες ελέγχου στις οποίες είναι η ίδια φυλακισμένη, έγκλειστη. Λοιπόν, υπευθυνοποίηση και απλούστευση είναι θα έλεγα δύο όψεις του ιδίου νομίσματος και από αυτές εξαρτώνται οι τάσεις αποτελεσματικότητας των περιφερειακών παρεμβάσεων, κάτι το οποίο επιθυμούν το σύνολο των εμπλεκομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου αναζητείται η ανάκαμψη και η έξοδος από την κρίση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ε, Thank you very much, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας σαν εκπροσώπου της οργάνωσής μου. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για ένα πολλά υποσχόμενο κείμενο εργασίας. Περιλαμβάνει ορισμένα σημεία τα οποία θα χαρακτήριζα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Θα σας εξηγήσω ακριβώς ε, σε τι αναφέρομαι. Πρώτον, η έκθεση αναφέρεται στη συνθήκη της Λισαβόνας σχετικά με τα προβλεπόμενα για τον σεβασμό των περιφερειακών και τοπικών αρχών όπως επίσης και την αρχή της επικουρικότητας. Οι αρχές αυτές θα πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως στην ολότητά τους. Έχουν χρησιμοποιηθεί στην προσπάθεια διατύπωσης της περιφερειακής πολιτικής και είναι πολύ θετικό για μας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει την εμπλοκή της σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ιδιαίτερα στην λεγόμενη προνομοθετική φάση. Είναι κρίσιμο να εμπλακούν οι περιφερειακές αρχές στη συζήτηση αυτή. Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές δεν είναι αυτοί που απλά εφαρμόζουν τις πολιτικές που καθορίζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εταιρική σχέση είναι ένα θέμα στο οποίο επιμένει πολύ η κυρία Μανέσκου και έχει δίκιο. Η βασική αρχή όμως αυτή της εταιρικής σχέσης θα πρέπει να εφαρμοστεί με τον σωστό τρόπο. Γι' αυτό άλλωστε και η εισηγήτρια ζητά και τα κράτη-μέλη και όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσουν σημασία στην σωστή εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης. Βασικός στόχος θα πρέπει να είναι για όλους και να συνεχίσει να είναι η συνοχή περιφερειακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα πρέπει να χαρακτηρίζει όλες τις ενέργειές μας και θα πρέπει να βρούμε τρόπους για να πετύχουμε τον στόχο αυτό. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για το μέλλον της περιφερειακής πολιτικής. Έχει σημασία επίσης και με τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Η εισηγήτρια ζητά να υπάρξει απλοποίηση των κανόνων και των διαδικασιών. Αυτό για μας είναι ένα κρίσιμο σημείο και θα πρέπει να υπογραμμιστεί ακόμα περισσότερο στην έκθεση Μανέσκου. Δυστυχώς η μέθοδος της χρηστής νομοθετικής ρύθμισης δεν είναι κάτι το οποίο έχει βοηθήσει μέχρι τώρα στην ελάφρυνση του γραφειοκρατικού βάρους, του γραφειοκρατικού άχθους. Το θέμα δεν είναι ε, μόνο η υπερβολική εργασία. Το πρόβλημα είναι ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές που έχουν ανάγκη από τα περιφερειακά ταμεία ουσιαστικά αποθαρρύνονται να ζητήσουν τα χρήματα αυτά λόγω της περιπλοκότητας των κανόνων. Τις ίδιες εμπειρίες έχω και από την πλευρά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εμπλεκομένων από την κοινωνία γενικότερα. Αυτό θα πρέπει να υπογραμμιστεί ακόμα περισσότερο στην έκθεση. Η συγγήτρια επιμένει ιδιαίτερα στα ελεγκτικά συστήματα της πολιτικής συνοχής. Η οργάνωσή μας προφανώς και πρέπει να είναι υπέρ του ελέγχου των δαπανών αυτών. Ταυτόχρονα όμως ανησυχεί διότι η εντατικοποίηση όλων των μορφών ελέγχων ορκωτών ημί είναι κάτι το οποίο δημιουργεί τελικά προβλήματα στη σωστή χρήση των ταμείων. Προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε και να υπακούσουμε στους κανονισμούς αυτούς, οι οποίοι όμως σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να βαίνουν περίπλοκοι και ακόμα περισσότερο στο μέλλον θα πρέπει να εφαρμόσουμε σωστά τις πολιτικές σύμφωνα με τους κανόνες που υπάρχουν και σύμφωνα με τους υπάρχοντες ελέγχους. Η έκθεση πάρα πολύ σωστά ζητά να υπάρξει μια πιο ενοποιημένη αντιμετώπιση όλων των ταμείων που έχουμε στη διάθεσή μας. Η σωστή χρήση των οικονομικών μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας έχει μεγάλη σημασία για να πετύχουμε πλήρως τους στόχους μας. Ενθαρρύνουμε την εισηγήτρια λοιπόν να υπογραμμίσει ακόμα περισσότερο το βασικό αυτό σημείο. Υποστηρίζουμε επίσης το αίτημα να εμπλέξουμε ακόμα περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συστήνουμε επίσης η έκθεση να δώσει τη δυνατότητα περισσότερης και μεγαλύτερης εμπλοκής των εκπροσώπων των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω τις εργασίες που έχουμε κάνει στον τομέα της πολιτικής συνοχής. Θεωρούμε ότι η πολιτική συνοχής έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έχουμε ήδη κυκλοφορήσει ένα κείμενο για τα βασικά πολιτικά μηνύματα της πολιτικής συνοχής. Έχω φέρει κάποια αντίγραφα της ε, εκθέσεως αυτής, του εγγράφου αυτού που έχει προετοιμάσει η οργάνωσή μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους για την ε, προσοχή. Ευχαριστούμε κύριε Γκούναρσον. Το λόγο κύριος Χέντριξ από το Σύνδεσμο Βιοτεχνιών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καταρχήν, εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιοτεχνιών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας και ιδιαίτερα την κυρία Μανέσκου για τη διοργάνωση αυτής της μήνυα ακρόαση και για την πρόσκληση μας εδώ. Καταρχήν, ποια είναι τα σχόλια μα ε, σε ό,τι αφορά τη Λευκή Βίβλο για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Μην ξεχνάτε ότι 92.500 τοπικές και περιφερειακές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλαμβάνουν πάνω από τα δύο τρίτα της Ευρωπαϊκής Ομοθεσίας. Είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή τους. Και μάλιστα η πλειοψηφία αυτών των νομοθετικών διατάξεων αφορά μέσα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η οικονομική και η κοινωνική πολιτική και οι βασικές προκλήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και η στρατηγική για το 2020, που είναι η δημογραφία, η ενέργεια, η παγκοσμιοποίηση, η απασχόληση, η βιώσιμη ανάπτυξη, ε, θα έχουν αντίκτυπο και στις βιοτεχνίες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλες αυτές οι πολιτικές λοιπόν θα πρέπει να εφαρμοστούν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο Αλλά μην ξεχνούμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, δεν μετεγκατίστανται και αποτελούν το 95% και το 55% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη δραστηριοποιούνται στην τοπική αγορά, στην εθνική αγορά και χρησιμοποιούν τοπική τεχνογνωσία. Γι' αυτό είναι σημαντική η περιφερειακή πολιτική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και το αντίστροφο. Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσει είναι σημαντικές για την περιφερειακή πολιτική. Σε ό,τι αφορά τώρα την πράσινη βίβλο για την δαφική συνοχή, ο σύνδεσμός μας τόνισε ότι τα επιτυχημένα περιφερειακά προγράμματα είχαν επιτυχία χάρη στο, στη σημαντική συνεργασία και ανάμειξη των τοπικών κοινοτήτων, των τοπικών επιχειρήσεων και των κοινωνικών εταίρων στις διάφορες περιφέρειες. Αντίθετα, σε εδάφη και περιφέρειες ε, όπου οι τοπικοί φορείς δεν συμμετείχαν στη διαβούλευση και εφαρμόστηκε ένα ενιαίο μοντέλο ανάπτυξης, ε, τα προγράμματα εκεί δεν είχαν τόσο μεγάλη επιτυχία. Οπότε το κλειδί της επιτυχίας των περιφερειακών προγραμμάτων έγκυται στην εταιρική σχέση μεταξύ των πολιτικών και των οικονομικών και κοινωνικών φορέων. Δηλαδή τη συνεργασία των πολιτικών αρχών με, τον, με τους κοινωνικούς και εταίρους και τους οικονομικούς τελεστές. Οπότε η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση θα πρέπει να λάβει υπόψη και την ανάγκη της πολυμορφίας των φορέων που συμμετέχουν σε αυτή τη διαβούλευση. Θα πρέπει συστηματικά να συμμετέχουν στην διαμόρφωση των προγραμμάτων που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις και που στόχο έχουν την εδαφική ανάπτυξη αλλά και την εφαρμογή των μεκών πολιτικών. Η επιτυχία της εταιρική σχέσης αυτής θα εξαρτηθεί από τρία κριτήρια. Καταρχήν την πολιτική βούληση για συνεργασία, δεύτερον την ανάγκη μια επιχειρησιακή νοοτροπία και κουλτούρα στη δημόσια διοίκηση και τρίτον οι εργασιακές μέθοδοι των προγραμμάτων, των προγραμμάτων θα πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επανέρχομαι στα τρία κριτήρια. Σίγουρα είναι επιτακτική ανάγκη τη πολιτική βούληση. Είναι αυτονόητο αυτό το κριτήριο, δεν χρειάζεται καν να αποδείξουμε την ανάγκη του. Επίση, ανάγκη επιχειρησιακή νοοτροπία τη δημόσια διοίκηση. γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αυτή η νοοτροπία στη δημόσια διοίκηση. Πολύ συχνά ε, είναι πολύ μονόπλευρη εντύπωση που έχει δημόσια διοίκηση για τις ε, επιχειρήσεις και ασχολείται περισσότερο με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ε, θα πρέπει οι διάφορες ε, πολιτικές να να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γιατί μια ομοιομορφοποίηση θα έχει αρνητικό αντικτύπο και για τις περιφέρειες αλλά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί οι πολιτικές δεν προσαρμόζονται στις διάφορες ιδιαιτερότητες και πραγματικότητες και στις μικρής κλίμακος επιχειρήσεις. Και επίσης ε, οι ενδιάμεσες οργανώσεις παίζουν ε, πολύτιμο ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ε, δημόσιων αρχών. Αυτός ο ρόλος δεν αναγνωρίζεται και δεν τη χάνει της δέουσας υποστήριξης ούτε από τις τοπικές ούτε από τις εθνικές διοικητικές αρχές. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι τα ευρωπαϊκά ε, περιφερειακά και δαφικά προγράμματα φτάνουν μέχρι τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μόνο όταν η εφαρμογή τους αναλαμβάνεται από διαμεσολαβητές, από ένα ενδιάμεσο επίπεδο δηλαδή διαχείρισης. Και φυσικά είναι ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι συγκεκριμένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα διάφορα προγράμματα. Σε ό,τι αφορά τις ανάγκες ελέγχου ε, και επιστοποίηση για τις μεγάλες επιχειρήσεις, η εφαρμογή ε, των επαχθέστατων γραφειοκρατικών διατυπώσεων αποκλείται de facto τι μικρομεσαίε επιχειρήσει από τέτοια προγράμματα θα πρέπει να αποφευθεί αυτή η υπερβολική γραφειοκρατία που επιβαρύνει ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στε, του στερεί την πρόσβαση στα κοινοτικά και περιφερειακά προγράμματα. Γι' αυτό και αποθαρρύνονται και χάνουν το ενδιαφέρον τους για τα διαρθρωτικά ταμεία. Σε ορισμένες περιφέρειες είχαμε εξαιρετικά αποτελέσματα αλλά μόνο 2 με 3% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι δικαιούχοι περιφερειακών προγραμμάτων και υποφελούνται μόνο σε επίπεδο 1-2% αυτών των διαρθρωτικών κονδυλίων, ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό και ο Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Βιοτεχνιών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων κατήρτισε ένα έγγραφο για την απλούστευση. Προτείνουμε 105 μέτρα απλούστευση των κανόνων σε ό,τι αφορά τους διοικητικούς κανόνες αλλά και την ε, δημοσιονομική διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων. Και τέλος κάποιες συστάσεις. Σύσταση πρώτη. Εφαρμογή των δύο βασικών αρχών ε, του, της πράξης για τις ε, μικρές επιχειρήσεις. Θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σημείο κλειδί της Λευκής Βίβλου είναι η γενίκευση της αρχής των, του Small Business Act σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Και μάλιστα συμμεριζόμαστε τη θέση της Λευκής Βίβλου που πιστεύει ότι η ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα περάσει από την ανάκαμψη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κάτι που προϋποθέτει εταιρική σχέση με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Όπως είπα και προηγουμένως, πάνω από το 95% όλων των επιχειρήσεων ενεργοποιούνται στις τοπικές αγορές. Συχνά όμως οι ευρωπαϊκές πολιτικές ε, χαράζονται και εφαρμόζονται για τις μεγάλες επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται δυστυχώς σε αντίθεση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παρόλο που οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι ένα τμήμα μόνο του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων. Γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που δημιουργούν περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Και μερικές φορές είναι αυτές που δίνουν το παρόν σε μειονεκτούσες περιοχές, ε, σε αστικές ζώνες ή σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές. Και ακριβώς επειδή βρίσκονται κοντά στον πολίτη θα πρέπει οι ανάγκες τους να ληφθούν υπόψη, με μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή. Θα πρέπει δηλαδή να ληφθούν οι ανάγκες τους σε τοπικό επίπεδο στα προγράμματα. Επίσης θα πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή του άπαξ και διαπαντός, σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά κονδύλια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε η αίτηση ε, και ο έλεγχος να πιστοποιείται από τις, εθνικές, από τις τοπικές αρχές χωρίς ανάγκη περαιτέρω ελέγχου και πιστοποίηση από τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές. Πρόκειται για ένα συμβολικό μέτρο για επιτυχούς και αποτελεσματικής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης θα ήταν η σύναψη μιας συμφωνίας μεταξύ των τριών θεσμικών επιπέδων της Επιτροπής Περιφερειών, και των τοπικών αρχών προκειμένου να περιοριστεί στο απολύτως απαραίτητο ο γραφειοκρατικός, το γραφειοκρατικό βάρος, οι διατυπώσεις ε, και η έλεγχη, εφαρμόζοντας την αρχή του, του άπαξ ελέγχου, που περιλαμβάνεται και στο Small Business Act. Επίσης, χρειαζόμαστε μια γενίκευση της νοοτροπίας του διαλόγου και μια οριζόντια επικουρικότητα η αρχή της οριζόντιας επικουρικότητας συνίσταται στην εξασφάλιση της συμμετοχής των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων στην διαδικασία της λήψης αποφάσεων και στη διαδικασία εφαρμογής των προγραμμάτων, όπως συμβαίνει με τη θεσμική και πολιτική επικουρικότητα. Σας ευχαριστούμε κύριε Χέντριξ. Έχουμε εδώ πρόσωπο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βλέπω εκπροσώπους και της Γενικής Διεύθυνσης ε, ε, περιφερειακής Ανάπτυξης, αλλά φαντάζομαι υπάρχει και εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας. Οπότε θα ήθελα αργότερα να ακούσουμε τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφού γίνει συζήτηση δηλαδή με τα μέλη της Επιτροπής. Ο Όντριχ Βλάσακ ζήτησε πρώτος το λόγο. Παρακαλώ, ποιοι άλλοι θέλουν να λάβουν μέρο στη συζήτηση για να προβλέψουμε μια δίκαιη κατανομή χρόνου. Όλτρι Βλάσακ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έγγραφο εργασία τη, που είναι πολύ σωστό βήμα προ την κατεύθυνση τη απλούστευση των κανόνων και τη καλύτερη χρήση των διαρθρωτικών κονδυλίων. Έχω πολλέ παρατηρήσει για την απλοποίηση των κανόνων. Αν θέλουμε να μα καταλαβαίνουν όλοι, θα πρέπει οι προτάσεις μας να είναι εύληπτες, απλές και κατανοητές. Μόνο έτσι θα μετα... μετατραπούν σε απτές λύσεις. Επίσης θα πρέπει να προσδιορίσουμε την εταιρική σχέση. Εταιρική σχέση σημαίνει δικαιώματα και υποχρεώσεις, αλλά ταυτόχρονα σημαίνει και μέθοδο για καλύτερη επεξεργασία αυτής της έννοια τη εταιρική σχέσης που χρήζει προσδιορισμό, όπω είπα. Και το μείζον θέμα της απλούστευσης. ρώτησε και τον αρμόδιο επίτροπο. Πώ εφαρμόζουν οι χώρες μέλη την αρχή της απλοποίησης, της απλούστευσης. Χρειαζόμαστε τέτοιες πληροφορίες για να κάνουμε μια σύγκριση μεταξύ των κρατών μελών. Για να δούμε τι κάνει η κάθε χώρα, ώστε να βοηθήσει στην απλοποίηση των κανόνων. Μιλήσατε για αυστηρότερο έλεγχο. Δεν κατάλαβα καλά. Τι εννοείται μεγαλύτερη πυγμή στον έλεγχο. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να ξέρουν οι εταίροι σαφώς και ξεκάθαρα ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους και τι έλεγχο να περιμένουν. Είμαι υπέρ του προγράμματος, της συνέχισης του προγράμματος ε, Έρασμος για τους τοπικούς και περιφερειακούς αντιπροσώπους. Και το θέμα της κατάρτισης είναι επίσης πολύ σημαντικό, γιατί θα πρέπει να επιμορφώσουμε τους συναδέλφους που είναι αρμόδιοι για τα θέματα ελέγχου. Επίσης, αυτό θα πρέπει να γίνει όχι μόνο σε συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών, αλλά πρώτα απ' όλα στη συνεργασία με τους Δήμους και κοινότητες των χωρών μελών. Γιατί αν είναι να διαλέξουμε τα κριτήρια της κατάρτισης ε, ή το ποιοι θέλουμε να υποφεληθούν από την κατάρτιση, αυτοί που έχουν αυτή τη γνώση είναι περισσότερο οι τοπικές και περιφερειακές αρχές. Επίσης, το θέμα των ε, διαφόρων μηχανισμών, θα ήθελα και το πρόγραμμα Jessica να περιληφθεί στα, στους μηχανισμούς του Financial Engineering. Ο κύριος Αγκουράκης. Αγκουράκης. Ε, vă mulțumesc, doamna președinte. Prefer să vorbesc pe românește pentru că sper că doamna Στα ρουμανικά, ο κύριος Αγκουράκη. σα ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω απευθείας ρουμανικά για να με καταλάβει καλύτερα, κυρία Μανέσκου. Νομίζω ότι θα πρέπει να διευκρινίσουμε καλύτερα το περιεχόμενο του εγγράφου εργασία της κυρίας Μανέσκου. Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν δύο βασικά προβλήματα εδώ. Η κυρία Μανέσκου προσεγγίζει το θέμα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση είναι ένα νέο θέμα και ένα νέο πρόβλημα και δημιουργεί έντονο προβληματισμό. Το έγγραφο εργασίας της κυρίας Μανέσκου δεν διευκρινίζει όλες αυτές τις απορίες που ανακύπτουν με το ζήτημα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Αναφέρθηκε το θέμα της συνεργασίας, για παράδειγμα, που και αυτό το θέμα θα πρέπει να προσδιοριστεί. Εγώ θα ασχοληθώ κυρίως με το δεύτερο τμήμα του εγγράφου, που αφορά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Μιλήσαμε εκτενώς για τα θέματα, για τα προβλήματα που υπάρχουν με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Και έχω πολλές απορίες, γιατί μιλούμε για πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Με μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση όμως δεν θα περιπλακεί και ο έλεγχος. Μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση δεν θα συνεπιφέρει και ένα πολυεπίπεδο έλεγχο. Γιατί η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση προποθέτει έναν κατακόρυφο άξονα και έναν οριζόντιο άξονα. Κάτι που απαιτεί όμως καλύτερο συντονισμό για να είναι θετικό το αποτέλεσμα. Οπότε, με όλες αυτές τις διαστάσεις και τα επίπεδα, περιπλέκεται και ο έλεγχος. Και όταν λέμε ότι θέλουμε απλούστευση του ελέγχου, τι εννοούμε. Μιλούμε, εννοούμε την ισχύουσα πρακτική που είναι ήδη αρκετά περίπλοκη και συμφωνώ ότι είναι περίπλοκη και χρήζει απλοποίησης. αλλά θέλουμε να εξασφαλίσουμε και μια αποτελεσματικότητα. Ή μήπως μας ενδιαφέρει μόνο η απλούστευση. Επίσης ε, φαίνεται το έγγραφο σαν πλήρως το πλαίσιο της οικονομικής κρίσης που σοβεί αυτή τη στιγμή και που βιώνουν όλες οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο η Ελλάδα ή η Ρουμανία. Διαρωτώ με λοιπόν πώς, ε, με ποιο τρόπο η ελληνική κυβέρνηση, η ουγγρική, η ρουμανική πώς θα χρηματοδοτήσουν τα μελλοντικά ευρωπαϊκά σχέδια και προγράμματα, ενώ αντιμετωπίζουν τεράστια δημοσιονομικά ελλείμματα. Ευχαριστώ. Thank you and Sean Kelly, please. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χέντριξ είπε ότι το 95% των επιχειρήσεων λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο και υπόκεινται σε κανόνες ε, οι οποίοι ισχύουν και για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι κάτι το οποίο επηρεάζει άμεσα και τη λειτουργία και την ίδια την κερδοφορία των μικρών επιχειρήσεων. Τι μπορεί να γίνει προς την κατεύθυνση αυτή λοιπόν. Ευχαριστώ. Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο. Ίσως ε, η ο κύριος Μάτουλα μάλλον έχει ζητήσει το λόγο, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ λοιπόν την <clears throat> κυρία Μανέσκου γιατί ασχολήθηκε με τα θέματα αυτά τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα εύκολα και δεν είναι σε καμία περίπτωση απλά θα ήθελα να επιμείνω στο θέμα της απλοποίησης των κανόνων, των κοινοτικών κανόνων αλλά και των εθνικών κανόνων φυσικά. Γιατί πρόκειται για μια εξαιρετική θα έλεγα ευκαιρία εδώ για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την τοπική διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα. Η απλοποίηση αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να λειτουργήσει μόνο σε, ε, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η απλοποίηση των κανόνων φυσικά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε θέματα ελέγχου. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε έναν πολιτισμό αξιολόγησης των επιδόσεων και στον τοπικό και περιφερειακό επίπεδο θα ήθελα παράλληλα να αναφερθώ και στις ε, δυνατότητες των μέσων Jeremy και Jaspers που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πλήρως και ελπίζω τα μέσα αυτά να χρησιμοποιηθούν καλύτερα. Καλώς συνάδελφοι, δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο. Θα ζητήσω λοιπόν από τους συναδέλφους της Αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κάνουν τα σχόλια τους. Η εμπειρία που έχουν και από την εφαρμογή των πολιτικών αυτών και από τις διαδικασίες ελέγχου, οι σχέσεις σαν παράδειγμα ελέγχου και αποτελεσματικότητας των πολιτικών μας. Τέτοιου είδους ε, σχέσεις και τέτοιου είδους κοινές μορφές διαχείρισης παρουσιάζουν προβλήματα Υπάρχει σωστή διαδραστική θα έλεγα συνεργασία. Τι γίνεται με τις δυνατότητες ελέγχου που έχει σε σχέση με τη διαχείριση του προϋπολογισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συνεχής αυτή σχέση που θα πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στον έλεγχο και την αποτελεσματικότητα. Σε ποια φάση βρίσκεται σήμερα, μπορείτε να μας μιλήσετε γι' αυτά. Άντερσον. Με χαρά. Θα σχολιάσω και εγώ το κείμενο εργασίας της κυρίας Μανέσκου. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω, παρουσιάζει πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες σχετικά με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαχειριστικών συστημάτων και της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών συστημάτων. Θα ήθελα επίσης να αντιδράσω σε ένα πρώτο επίπεδο στο έγγραφο αυτό, να υπογραμμίσω το τι κάνουμε και τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα για τη βελτίωση των ελεγκτικών συστημάτων. Βλέπουμε με ικανοποίηση ότι γίνεται θετική αναφορά στο πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον ελεγκτικό της ρόλο. Τα πρώτα αποτελέσματα που έχουμε από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, από το παρόν πρόγραμμα φαίνονται θετικά και ε, με χαρά θα ήθελα να έρθουμε σε στενότερη επαφή με την εισηγήτρια και την ομάδα της για να μοιράσουμε μεταξύ μας περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες. Έχουμε λοιπόν ένα νέο νομικό πλαίσιο σε αυτή τη βάση, μια νέα νομική βάση. Έχουμε ενισχύσει το ρόλο των εθνικών και περιφερειακών ελεγκτικών αρχών και όπως έλεγε και η συγγήτρια έχουν υπάρξει ερωτηματικά σε σχέση με την πιθανότητα επικαλύψεων και κακού συντονισμού των διαδικασιών ελέγχου. Αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα αντιμετωπιστεί έτσι ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε βασιζόμενοι στα αποτελέσματα των εθνικών μορφών ελέγχου έχει μεγάλη σημασία για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε σωστά τα νέα αυτά προγράμματα που έχουμε μπροστά μας. Είμαστε στην αρχή της προγραμματικής περίοδου, αυτό υπογραμμίζεται έτσι και αλλιώς άλλωστε στο έγγραφο Μανέσκου. Έχουμε επίσης And also we are providing guidance on the first uh, level control provisions to... Έχουμε επίσης ε, ασχοληθεί με το θέμα της ε, συμβατότητας ε, των δηλώσεων συμβατότητας μάλλον των προγραμμάτων αυτών σε σχέση με τις απαιτήσει οι οποίες έχουν διαμορφωθεί τις λεγόμενες δηλώσεις συμμόρφωσης. Έχουμε οργανώσει επίσης ε, τα σεμινάρια εκπαίδευσης των εκπαιδευτών. Έχουμε κάνει παρουσιάσεις, εργαστήρια στις τοπικές αρχές, στις περιφερειακές αρχές, έτσι ώστε και αυτές με τη σειρά τους να οργανώσουν σεμινάρια άμεσα για τους εμπλεκομένους. Για τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα και τις μορφές ελέγχου. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα είναι να αποφύγουμε τις επικαλύψεις με τους ελέγχους και θα πρέπει να θεωρούμε αξιόπιστες τις ελεγκτικές διαδικασίες των τοπικών και εθνικών αρχών. Το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Έχουμε προωθήσει και διαφορετικές δράσεις στα πλαίσια της κοινή ελεγκτικής διαδικασίας, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία επικαιροποίηση. Δηλαδή εμείς ελέγχουμε όλες τις υπηρεσίες των διαφορετικών ταμείων και όταν ολοκληρώσουμε τον έλεγχο αυτό σε λίγες εβδομάδες, τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα τα στείλουμε και στη δική σας επιτροπή, έτσι ώστε <clears throat> να μπορέσετε να εκφράσετε και εσείς τις δικές σας απόψεις. Ένα άλλο θέμα είναι το επίκαιρο του συγκεκριμένου εγγράφου, έτσι ώστε να έχουμε σαφέστατα στη διάθεσή μας τα απαιτούμενα μέσα για την περίοδο μετά το 2013 και εδώ η εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι απόλυτα θετική. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Υπάρχουν και ερωτηματικά σχετικά με αυτά τα οποία έλεγαν οι συνάδελφοι που δεν έχουν απαντηθεί κυρία Μανέσκου, σαν παράδειγμα αυτά που είπε ο Σον Κέλλη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. <coughs> Ίσως να μην κατάλαβα την ερώτηση του κυρίου Κέλλη. Είπα πράγματι ότι το 95% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο μόνον και αυτό δεν θα πρέπει να συγχαίεται με την, με την κερδοφορία τους και την αποδοτικότητά τους. Τι μπορούν να κάνουν ε, για να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Αυτή ήταν η ερώτησή σας κύριε Κέλλη. Όχι, όχι. Υπόκεινται σε κανόνες και νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες ισχύουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουν σχεδιαστεί για μεγάλες επιχειρήσεις διεθνικές. Υπόκεινται λοιπόν σε διαδικασίες οι οποίες δεν είναι απαραίτητες για το δικό τους επίπεδο λειτουργίας. Πράγματι. Το πρόβλημα είναι, λέει ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας συλλαμβάνεται, αν θέλετε, και διαμορφώνεται για τις μεγάλες ε, επιχειρήσεις, ε, για τις διεθνικές επιχειρήσεις, και είναι αλήθεια ότι αυτοί που σχεδιάζουν τις νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις δεν ασχολούνται με τις μικρομεσαίες και τις μικρές επιχειρήσεις. Η, η μικρή επιχείρηση δεν είναι βέβαια κάτι το οποίο λειτουργεί ε, σε μικρότερο επίπεδο ε, με τον τρόπο λειτουργίας μιας μεγάλης επιχείρησης. Περισσότερο ισχύει το αντίθετο βέβαια. δεν λαμβάνονται υπόψη, δεν λαμβάνονται υπόψη οι, μικρές, ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις απαραίτητα στη διαμόρφωση των νομοθετικών ρυθμίσεων. Και αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι ακριβώς να εξηγήσουμε στους πολιτικούς και στους νομοθέτες πώς λειτουργεί μια μικρή επιχείρηση, μια μικρομεσαία επιχείρηση. Ελπίζω αυτό να απαντά την ερώτησή σας. Ξέρει την απάντηση στο ερώτημα αυτό ο Σον Κέλλη βέβαια, είναι ικανοποιημένος από αυτά που είπατε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω δύο ακόμα λόγια σε ό,τι αφορά την απλούστευση, παρότι ε, αποτέλεσε ένα από τα κύρια σημεία στα οποία εστίασε αυτή η συζήτηση. Εγώ ανησυχώ πολύ ε, σήμερα για τα διαρθρωτικά ε, ταμεία ε, και αυτό γιατί εγώ προεδρεύω σε μία από τις εταιρικέ σχέσεις της Σουηδία η οποία έχει ε, χωριστεί σε 8 εταιρικέ σχέσεις και σας λέω σε μία από αυτές προεδρεύω εγώ. Στη δική μας λοιπόν περιφέρεια έχουμε 52 δήμους και κοινότητες και όταν κάνουμε συζητήσεις με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα σε αυτήν την δική μας περιφέρεια πολλοί προσωποί μας λένε όχι δεν θα υποβάλουμε αίτηση για χρηματοδότηση από το Διευθυντικό Ταμείο γιατί είναι υπερβολικά περίπλοκη η διαδικασία. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ χρόνο για να συντάξουμε μια αίτηση και από εκεί και μετά ο μηχανισμός ελέγχου και εποπτείας είναι πολύ δύσκολος. Και μιλάμε για τοπικούς και, τοπικές και περιφερειακές αρχές. Όταν κάνουμε ε, συζητήσεις τώρα με μικρές επιχειρήσεις για χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία μας λένε πως είναι πολύ δύσκολη διαδικασία, πολύ περίπλοκη για να ε, γίνει ε, τόσο σε ό,τι αφορά το επίπεδο της υποβολής μιας αίτησης αλλά και σε ό,τι αφορά το επίπεδο του ελέγχου. Και με ανησυχεί πολύ αυτό γιατί το Ταμείο αποτελεί ένα ορατό παράδειγμα αλληλεγγύης στην Ευρώπη και ένα παράδειγμα ε, σε ό,τι αφορά την παρουσία της Ευρώπης στην ίδια τη Σουηδία. Άρα λοιπόν, αν εμείς αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα στη Σουηδία, σίγουρα και εσείς αντιμετωπίζετε πολλά αντίστοιχα τέτοια προβλήματα στις ε, πατρίδες σας. Ε, αυτό αποτελεί πρόβλημα επειδή με τη χρήση των ταμείων μπορεί κανείς να αξιοποιήσει, να κινητοποιήσει αν θέλετε κονδύλια από διαφορετικούς φορείς στην κοινωνία, ώστε να προωθήσει την ανάπτυξη και της, της εν λόγω Άρα λοιπόν είναι κέρια σημασίας αυτό το ζήτημα. Πώς να καταστεί αυτή η διαδικασία ε, αν θέλετε υποβολής αίτησης και ελέγχου στο πλαίσιο της χρηματοδότησης των ε, διαρθρωτικών ταμείων. Ε, και ένα ακόμα ζήτημα είναι ότι δεν έχει κανείς αρκετά κονδύλια εκ των προτέρων. Δηλαδή για να λάβει κανείς μια χρηματοδότηση, αν θέλετε, περνάνε εννέα μήνες. και για να μπορεί κανένα να, να περιμένει για τόσο καιρό σημαίνει ότι ήδη είναι αρκετά ισχυρό ε, για να μπορέσει λοιπόν να υποβάλει μια αίτηση για το ε, για χρηματοδότηση από διευθυντικά ταμεία ε, και καλό θα είναι να εστιάσει αυτή η έκθεση ε, σε, σε αυτά τα αισθήματα. Ναι, ε, Πρόεδρος, ε, νομίζω πως υπάρχει αυτή, η πολύ δυνατή σχέση μεταξύ good governance και της διακυβέρνησης και της διαχείρισης. Θέλετε να πάρετε ξανά τον λόγο για να σχολιάσετε, δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, τους εμπειρογνώμονές μας προσκεκλημένους που έλαβαν το λόγο, τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ για τις ε, συστάσεις και τις παρατηρήσεις που έκαναν και είμαι πεπισμένη ότι η έκθεσή μου θα εμπλουτιστεί και θα βελτιωθεί, θα βελτιωθεί χάρη στη συνεργασία μεταξύ μας και στην ανάγκη να υλοποιήσουμε τους κοινούς μας στόχους. Όλοι θέλουμε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των δικαιούχων στα διαρθρωτικά κονδύλια. Αυτό είναι ο πρωτερχικός μας στόχος. Και αυτό θα το καταφέρουμε μέσω της εταιρική σχέσης, της επιμόρφωσης, της απλοποίησης. Απλοποίηση προϋποθέτει και μεγαλύτερη συνδρομή προς τους δικαιούχους, ώστε να μειωθεί το περιθώριο λάθους και των παρατυπιών. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, πολλές φορές έχουν γίνει απλουστεύσεις των κανόνων. Αλλά ο τρόπος που μεταφέρθηκε η απλοποίηση αυτή σε εθνικό επίπεδο ήταν πολύ διαφορετικός από χώρα σε χώρα. Και υπάρχουν δυσκολίες με την πρόσβαση στα κονδύλια στις διάφορες χώρες. Εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως το συμφέρον των δικαιούχων και το πώς θα εξασφαλιστεί ευκολότερη πρόσβασή τους στα διαρθρωτικά κονδύλια. Αν έχουμε κατά νου τους δικαιούχους, θα καταφέρουμε να συνδράμουμε και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές για να εξασφαλίσουν διευκόλυνση της πρόσβασης στα διαρθρωτικά κονδύλια. Σας ευχαριστώ θερμά και περιμένω και γραπτός τις προτάσεις για την έκθεσή μου. Thank you ε, very much. Thanks to, to everybody. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους που συμμετείχαν στην σημαντική αυτή συζήτηση για την πολύ σημαντική έκθεση. Θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία, γιατί είναι πολλές οι προκλήσεις που συνδέονται με αυτό το είδος επίπεδης διακυβέρνησης. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε και τα χρήματα των φορολογουμένων, να αξιοποιήσουμε τον κοινοτικό προϋπολογισμό, να αυξήσουμε τις θέσεις απασχόλησης, αλλά ταυτόχρονα να μην επιδεινώσουμε το γραφειοκρατικό άχθος. Και ήταν η πρώτη φορά σήμερα που ακούσαμε ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια να συνδυάσουμε όλους αυτούς τους παράγοντες και να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ τόσο διαφορετικών προκλήσεων, θα πρέπει ως σημείο αναφορά μας να έχουμε τον τελικό αποδέκτη, τον δικαιούχο των ε, διαρθρωτικών ταμείων. Καλό θα ήταν λοιπόν όταν προσεγγίζουμε την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση να έχουμε ένα συγκεκριμένο πρίσμα. Αυτό είναι κάτι που ακούσαμε σήμερα. Μήπως θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα, όπως είπατε εσείς, ε, στο συμφέρον του δικαιούχου και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία να υποτάσσονται σε αυτό τον πρωταρχικό στόχο που είναι το συμφέρον του δικαιούχου. Ή να προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε τους διάφορους παράγοντες και να βρούμε μια σωστή ισορροπία υπό ποιο πρίσμα θα προσεγγίζουμε την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, υπό το πρίσμα του συμφέροντος του δικαιούχου ή υπό το πρίσμα της ανέβρεσης ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων προκλήσεων. Πολύ ενδιαφέρον πάντως το σχόλιο σας. Και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή συνάδελφοι σε μια λέξη που ακούσαμε από τις ομιλίες και που ήταν το θέμα της σύμβασης του συμβατικού χαρακτήρα, να έχουμε συμβατικού είδους συμφωνίες για, τη, για τα περιφερειακά προγράμματα μεταξύ των δικαιούχων, των τοπικών και περιφερειακών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η ιδέα του συμβολέου ακούστηκε πολλές φορές. Περιμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες και εξηγήσει για αυτή την προσέγγιση, γιατί εμφανίζεται πια το θέμα Τη σύμβαση, του συμβολέου και του συμβατικού χαρακτήρα της προσέγγισης σε πολλά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είπατε ότι θα μπορούσε να είναι και ένα μέσο για την απλούστευση των κανόνων αυτός ο συμβατικός χαρακτήρας. Περιμένουμε λοιπόν πιο διεξοδικές προτάσεις για το μέλλον της της πολιτικής αυτής. Αυτά και ολοκληρώσουμε το συγκεκριμένο σημείο της σημερινής διάταξης. Ευχαριστώ θερμά πάλι τους καλεσμένους.